Äh, Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Δεν είμαστε ακόμα όλοι παρόντες. Η Επίτροπος ήρθε νωρίς, διότι αύριο έχει να πάει στην Κίνα. Και σας ευχαριστώ που κάνατε τον κόπο να έρθετε. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή γιατί όλοι έχουμε ε, λιγάκι υποστεί κάποια σύγχυση λόγω των προτάσεων οι οποίες υπάρχουν και θα θέλαμε ε, να ξέρουμε πώς το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόκειται να εφαρμοστεί. Δηλαδή θα έπρεπε ε, να σας πούμε να μπορούμε να σας πούμε πού χρησιμοποιεί κανείς ε, την λανθασμένη οδό. Οπότε, σας ευχαριστώ που ήρθατε κυρία Βασιλείου. Μήπως μπορείτε καταρχήν, πρώτα απ' όλα, ε, ημερήσια διάταξη. Φαντάζομαι ότι κανείς δεν έχει τίποτα κατά της ημερησίας διατάξεως. Μετά προχωράμε στα πρακτικά της προηγούμενης συνεδριάσεως. Αν μέχρι το βράδυ δεν έχει υπάρξει καμία αντίρρηση για το πρακτικά θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί. Διαφορετικά παρακαλώ να μου υποβάλλετε τις προτάσεις σας για αλλαγές. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίαση αυτή ε, και πάλι ε, εκπέμπεται και γι' αυτό ε, δεν μ' αρέσει να έχουμε τόσες άδειε θέσεις μπροστά μπροστά. Θα ήθελα να σας πω ότι ορισμένες γλώσσες δεν μεταφράζονται ε, εστονικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα Σλοβάκικα, Βουλγάρικα και Σουηδικά δεν υπάρχουν, όλες οι άλλες γλώσσες μεταφράζονται. Εάν θέλετε όμως να μπορείτε να μιλήσετε Ολλανδικά και Πορτογαλικά και από τις γλώσσες αυτές υπάρχει μετάφραση, όχι όμως προς τις γλώσσες αυτές. Ωραία, αύριο έχουμε δύο ψηφοφορίες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αύριο έχουμε ψηφοφορίες και να φέρετε μαζί σας τις ε, κάρτες σας ψηφοφορίας διότι καλό θα ήταν να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τις εκθέσεις Βαντία και ε, ναι, Ντάλοβα. Τώρα λοιπόν έχουμε τη συζήτηση με την Επίτροπο. Χαίρομαι ιδιαίτερος που είστε εδώ σήμερα και θα ήθελα να μας παρουσιάσετε την ημερήσια διάταξη αυτού του έτους ή και λιγάκι τα θέματα για το επόμενο έτος γιατί δεν θα έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά εντός του έτους. Σας δίνω το λόγο για να συζητήσουμε όλοι μαζί αυτά τα θέματα. Κυρία Βασιλείου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή είναι η πρώτη μου επαφή μαζί σας από όταν ε, ανέλαβα καθήκοντα και έχουμε μία πολύ πλούσια ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα λοιπόν πολύ να μπορέσω προτού ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα εργασίας μας, να ακούσω τις προτάσεις σας και να τις συζητήσω μαζί σας. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι όσο περισσότερο Υπησέρχομαι στα θέματα της αρμοδιότητός μου, τόσο περισσότερο βλέπω ότι όλα τα θέματα τα οποία χειρίζομαι επηρεάζουν άμεσα τους ανθρώπους τους πολίτες και το βλέπω όταν συναντώ τα παιδιά, τους φοιτητές του προγράμματος Έρασμος, ε, το πρόγραμμα ε, τους νέους εκπροσώπους εις το Φόρουμ Νεολαία στη Χερέθ και επιπλέον, και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, πολλοί από τα άτομα με τα οποία συναλλασσόμαστε είναι νέοι. Νέοι ε, οι οποίοι διαμορφώνονται για την επόμενη δέκα δεκαετία που είναι το αντικείμενο του προγράμματος παρουσίασε τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος Μπαρόσο. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι όλοι ενδιαφερόμαστε πολύ για τις πολιτικές μας. Ο στόχος μας είναι Ευρώπη του 2020, δηλαδή η στρατηγική μας για μια φόρα έξυπνη και γενική ε, παιδεία. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι ε, κοινωνία θέλει η Ευρώπη όταν θα εξέλθει από την κρίση. Και αν πιστεύουμε ότι θέλουμε ε, να έχουμε σαν κλειδί για το μέλλον την ισότητα, ε, τότε θα πρέπει η εκπαίδευση να είναι στο επίκεντρο της κοινωνίας και να εξασφαλίσει ότι όλοι θα μπορέσουν να αποφαληθούν. Στηρίζεται η παιδεία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και κάμποσο κελό. Η Ευρώπη του 2020 ανανεώνει αυτή την υποχρέωση και τη δέσμευση και η στρατηγική αποδεικνύει ότι η εκπαίδευσή μας και τα ερευνητικά κέντρα θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να ε, αναδιαμορφώσουμε ε, μια συνολική και έξυπνη ανάπτυξη. Βλέπω στενούς δεσμούς μεταξύ της Ευρώπης 2020 ε, και του πλαισίου για την συνεργασία στην Ευρώπη στον τομέα της παιδείας και της επιμορφώσεως και προσβλέπω στην ανάγνωση της εκθέσεως την οποία καταρτίζει η κυρία Μπαντία. Πιστεύουμε ότι μέχρι το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή πιστεύει ότι όλοι ε, ε, τα παιδιά τα οποία φεύγουν νωρίς από το σχολείο θα έχουν μειωθεί κάτω του 10% θα είναι απόφατοι της ανωτάτης εκπαιδεύσεως ή αντιστοίχου. Ε, θα ήθελα λοιπόν να διορθώσω και να τονίσω ότι μιλάμε για την πανεπιστημιακή ή ισότιμη εκπαίδευση. Εάν λοιπόν ε, ε, ε, θέλουμε οι στόχοι αυτοί να γίνουν πιστευτοί, θα πρέπει όλοι να εξασφαλίσουμε ότι οι νέοι θα ξεκινήσουν κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν να έχουν τα εχέγγυα για να ε, διαμορφώσουν έναν πλήρη και δραστήριο ρόλο στον κόσμο. Έχουμε ε, τέσσερα ε, βασικά μηνύματα. Νεολαία εγκινήσει, νέες δεξιότητες και απασχολήσεις, η ένωση της καινοτομίας και η ψηφιακή ατζέντα. Θα αναφερθώ και θα σχολιάσω κάθε ένα από αυτά τα θέματα και για να το κατανοήσετε. Λοιπόν, όσον αφορά την νεότητα εν κινήσει, η κρίση έχει χτυπήσει πάρα πολύ τους νέους Ευρωπαίους και η ανεργία των νέων είναι γύρω στο 20%. Πήγα στην Ισπανία και είδα ότι εκεί η ανεργία των νέων φτάνει στο 39%. Η κατάσταση δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημη. Άρα το πρόβλημα των νέων της Ευρώπης είναι πρόβλημα ολόκληρης της Ευρώπης και δεν μπορούμε να χάσουμε ε, χρόνο ή να σπαταλήσουμε αυτά τα ταλέντα. Και γι' αυτό πρέπει να βελτιώσουμε την παιδεία, το οποίο ήδη αποτελεί μία σημαντική πρόκληση. Χρειαζόμαστε να ξανασκεφτούμε τη σχέση της παιδείας με την υπόλοιπη κοινωνία κοινωνία, να βρούμε νέους τρόπους να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες στην Ευρώπη για την καινοτομία και γι' αυτό χρειαζόμαστε την νεολαία εγκινήση. Πράγμα το οποίο θα περιλάβει και ένα νέο πλαίσιο πολιτικής και ένα νέο πρόγραμμα. Σκοπεύω να παρουσιάσω το πλαίσιο της πολιτικής σε μία ανακοίνωση τον Ιούνιο, ενώ οι προτάσεις για ένα νέο πρόγραμμα θα ε, παρουσιαστούν μόνο του χρόνου. Η νεολαία εγκινήση θα συγκεντρώσει και θα συνδυάσει σε όλες υπάρχουσες προσπάθειες και θα τις διοχετεύσει σε τέσσερις ε, τομείς. Δηλαδή θα προωθήσουμε την αριστεία στην ανωτάτη εκπαίδευση, την κινητικότητα σε όλες τις βαθμίδες εκπαιδεύσεως, ένα σύγχρονο σύστημα διαβίου μαθήσεως και την απασχόληση των νέων και τη συμμετοχή των νέων. Όσον αφορά την αριστεία, πιστεύω ότι μπορούν τα πανεπιστήμια μας να έρθουν πιο κοντά στην κοινωνία χωρίς να υπονομεύσουμε την αυτονομία τους. Η, τα πανεπιστήμια παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο πέραν της παιδείας και της έρευνας στόχος μας είναι να προσαρμόσουμε τις ε, καλύτερες προοπτικές της Ευρώπης στις ανάγκες ενός ε, κόσμου εν εξελίξη. Το περασμένο μήνα το, ε, η επέτειος της διαδικασίας της Μπολόνια ξεκίνησε ε, επισήμως στον τομέα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανωτά της Εκπαιδεύσεως το γεγονός αυτό ήταν μια επιτυχία και εξασφαλίζουμε ε, ότι θα επιτρέψουν οι πανεπιστημιακές δεξιότητες στους νέους να ε, φτάσουν στην ανώτατη δυνατή ποιότητα και να προετοιμαστούν για την ε, οικονομία της γνώσεως τα εκπαιδευτικά μας συστήματα πρέπει να αντιδρούν καλύτερα στις αλλαγές της κοινωνίας, να προωθήσουν τη δυνατότητα απασχολήσεως των φοιτητών και ε, να προωθήσουμε τις στενές συνεργασίες μεταξύ ε, ε, των επιχειρήσεων και της παιδείας και θέλω να συγχαρώ τον Πάουλ Σμιτ για την έκθεσή του όσον αφορά το διάλογο μεταξύ πανεπιστημίου και επιχειρήσεων. Ε, θεωρώ ότι αυτό συνεχίζει την εργασία την οποία ξεκινήσαμε και ε, πιστεύω ότι πρέπει να ε, ε, διατηρήσουμε την αυτονομία των πανεπιστημίων αλλά και να προωθήσουμε τη συνεργασία. Συγχρόνως η διαφάνεια των θεσμών ανωτά της εκπαίδευσης είναι πολύ βασική, να, μπορούν δηλαδή οι φοιτητέ να κάνουν εν πλήρη γνώση τις επιλογές τους και θέλω να σκεφτώ ότι ε, θα μπορέσουν όλοι οι νέοι να υποφεληθούν από την ανώτατη εκπαίδευση κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν να έχουν έχουν επικερδεί και ικανοποιητική εργασία. Η πρόθεση της κινητικότητας είναι ο δεύτερος στόχος ε, του προγράμματος της ε, ε, νεολαίας εν κινήσει. Η κινητικότητα είναι μεγάλη επιτυχία ή στην ευρωπαϊκή παιδεία, σκεφτείτε τον Κομένιο, στον Έρασμο και τη Μαρή Κιουρί. Ε, και ε, κατά αυτόν τον τρόπο η κινητικότητα διευρύνει τους ορίζοντες αλλά ε, η κινητικότητα πρέπει να ισχύει για όλους τους νέους και όχι μόνο για τους φοιτητές και τους ερευνητές. Η κινητικότητα δεν μπορεί να είναι μόνο μία πολυτέλεια μιας μικρής εξέχουσας τάξεως, αλλά να μπορεί να συμπεριληφθεί για κάθε νέο Ευρωπαίο. Και τώρα με πολύ ισχυρές δράσεις όπως το πρόγραμμα Έρασμος μπορούμε να προσεγγίσουμε μόνο ένα μικρό ποσοστό των φοιτητών ενώ θεωρούμε ότι οι δράσεις κινητικότητας σε όλους τους τομείς της παιδείας θα πρέπει να μπορέσουν ε, να ε, διατεθούν σε 370.000 νέους ετησίως. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και θα πρέπει να ε, καταργήσουμε τα διάφορα προσκόμματα στην κινητικότητα για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ε, θα πρέπει να δοθεί η οικονομική στήριξη στους φοιτητές και να αναγνωριστεί η ε, επίσημη, άτυπη και ανεπίσημη ε, παιδεία και εκπαίδευση η οποία αποκτήθηκε στο εξωτερικό. Θα πρέπει δηλαδή να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε ε, αυτούς που μειονεκτούν να έχουν τις ίδιες ε, δυνατότητες με όλους και να διευρύνουμε τις ομάδες που πηγαίνουν παραδοσιακά στο πανεπιστήμιο. Η ε, κοινωνία της γνώσης χρειάζεται τα ταλέντα όλων και πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερη κινητικότητα ε, για τους εκπαιδευόμενους και τους εθελοντές και το νέο πρόγραμμα Κομένιους είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση Ελπίζουμε δε ότι έτσι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μία πιο μακροπρόθεσμη κινητικότητα και για τους διδάσκοντες. Όσον αφορά ε, τα συστήματα ε, της ε, αηφόρου μάθησης, της διαβίου μάθησης, και την κατάρτισή τους θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μέχρι το 2020 ότι 50% των θέσεων εργασίας θα εξαρτώνται από τις δεξιότητες μέσης εκπαίδευσης που προσφέρει η επαγγελματική κατάρτιση. Θα πρέπει όμως να την εξυγχρονίσουμε διότι σε πολλές χώρες η εικόνα της επαγγελματικής κατάστασης δεν κατάρτισης δεν είναι καλή ε, για τους νέους και θα πρέπει να ενταχθούμε από τις αλλαγές της αγοράς εργασίας και να δούμε τι λειτουργεί καλύτερα στα κράτη-μέλη και ε, να μπορέσουμε από τους εκπαιδευόμενους ε, ε, να μάθουμε και να τους προσφέρουμε μεγαλύτερη κινητικότητα για να διδαχθούν. Να ξαναξεκινήσουμε και τη διαδικασία της Κοπενχάγης και σκοπεύω σύντομα να παρουσιάσω μία ανακοίνωση στους συναδέλφους μου για την επαγγελματική πολιτική που να στηρίζουν τους στόχους της στρατηγικής του 2020. Θα ήθελα επίσης να εστιαστώ στο δύσκολο πρόβλημα της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου που είναι μια μεγάλη αδυναμία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εκπαιδεύσεως και χάσιμο χρόνου. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να μπορέσουν οι νέοι μας να έχουν επαρκή παιδεία και να ενισχύσουμε την αντοχή τους και να τους βοηθήσουμε στις τις διαδικασίες της εκμάθησης. Γι' αυτό και είναι βασικό να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους διδάσκοντες και το εκπαιδευτικό προσωπικό που φροντίζουν τα παιδιά μας. Θα πρέπει επίσης να ασχοληθούμε με την πρόληψη, δηλαδή να βρούμε τρόπους με τους οποίους να βρούμε ποιοι είναι οι επικίνδυνοι ε, μαθητές οι οποίοι θα εγκαταλείψουν το σχολείο ή αν εγκαταλείψουν το σχολείο να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία και να τους δώσουμε νέες δυνατότητες για να επανέλθουν στο ε, σύστημα το εκπαιδευτικό διότι η ε, νεολαία κινήση δεν αναφέρεται μόνο στην νεολαία. Αναφέρεται σε όλη μας την εργασία και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν ε, ε, ιδιάζον σύνολο προβλημάτων να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουν να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία και να εκφράσουν όλες τις δυνατότητές τους. Και αυτός είναι ο τέταρτος και τελικός στόχος του προγράμματος Νεολαία Εγκινήση. Ε, θέλω να χαιρετήσω το ενδιαφέρον της Επιτροπής σας για τη στρατηγική νεολαία. Θέλω να χαιρετήσω την έκθεση Παπα-Νικολάου και το ότι τονίζει την κοινωνική ένταξη των παιδιών των μεταναστών. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί με την ανεργία και γι' αυτό θα συνεργαστώ στενά με τον συνάδελφό μου Επίτροπο Άντορ και μέχρι το τέλος του χρόνου θα προτείνουμε μία ανακοίνωση σε ένα νέο πλαίσιο απασχολήσεως της νεολαίας για να υπάρχει μία πιο ομαλή μετάβαση από την ε, εκπαίδευση ή στην αγορά εργασίας. Θα περιλάβουμε επίσης ε, στην Ευρωπαϊκή ε, Στρατηγική Απασχόληση τα στοιχεία αυτά και θα τα προωθήσουμε για να ε, διαθεθούν και οι ευρωπαϊκοί πόροι οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην κρίση, ιδίως στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ε, έχουμε όμως ε, και άλλα συνθήματα για το, τη στρατηγική του 2020 ε, που αναφέρονται καταρχήν στην καινοτόμα ένωση. Δηλαδή πρέπει να ενισχυθούμε για να αντεπεξέλθουμε από την κρίση και ε, να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες διότι έχει επιταχυνθεί ε, η ε, αλλαγή στην κοινωνία μας και όσο αλλάζει η κοινωνία αλλάζει και η εργασία. Υπάρχουν ορισμένες εργασίες που καταργούνται, άλλες οι οποίες προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες στην πράσινη οικονομία ή στην υγεία και στον τομέα της περίθαλψης διότι έχουμε ένα γυράσκοντα πληθυσμό αλλάζουν και τα μέσα και οι δυνατότητες. Οι τεχνικές γνώσεις θα είναι πάντοτε αναγκαίες, αλλά συγχρόνως είναι σημαντικό να υπάρχουν οι δεξιότητες που θα επιτρέψουν στους νέους να αποκτήσουν νέες γνώσεις. Χρειαζόμαστε τη δεξιότητα της καινοτομίας και με την, το πρόγραμμά μας των νέων δεξιοτήτων και καινοτομιών θα προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τις δυνατότητες απασχολήσεως ε, για ε, τις επιχειρήσεις και για όλους τους κοινωνικού εταίρους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες και θα αναφέρω ορισμένες ιδέες. Προσπαθούμε να υπάρξει μία κοινή γλώσσα για να ε, ε, εξηγήσουμε τις δεξιότητες και τις εργασίες κατά τρόπον ώστε να βελτιωθεί η ανάλυση της αιτήσεως για δεξιότητες και να στηρίξει την δυνατότητα ε, βοηθείας προς τους εργοδότες ε, και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Θέλουμε να ταιριάξουμε ε, τις εργασίες με την τεχνολογία, αλλά η γνώση δεν είναι αυτός σκοπός, οπότε θα πρέπει να υπάρξουν ευρωπαϊκά ε, συμβούλια δεξιοτήτων, όπου ο καθένας να μπορεί να υποφελείται από τις ιδέες κάποιου άλλου. Ε, φίλοι μου, επιτρέψτε μου τώρα να αναφέρω ποια είναι τα άλλα δύο θέματα της ε, ε, Ευρώπης του 2020. Αύριο θα δημιουργήσω δύο, ένα, ε, ε, αύριο θα δημοσιεύσω ένα νέο έγγραφο σχετικά με την καινοτόμα ένωση για να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών για να μπορέσουν όλοι να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες τους και θα έπρεπε επίσης να αναφέρω το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας που τώρα έχει καταρτήσει τις τρεις πρώτες κοινωνίες καινοτομίας που θα αρχίσουν να εργάζονται σύντομα συμβάλλω και σε ένα τελικό θέμα που είναι η ψηφιακή ατζέντα. Δηλαδή οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν διευρύνει την πρόσβαση στο δημιουργικό περιεχόμενο και θέλουμε να διατηρήσουμε την ε, δημιουργική και πολιτιστική πολυμορφία. Και επικεντρωνόμαστε σε τρεις τομείς, ε, την πνευματική ιδιοτηξία, την ψηφιακή ε, ε, την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στους κινηματογράφους και ε, την ψηφιακή ε, χρήση πολιτιστικού περιεχομένου. Θα συνεργαστώ στενά με την κυρία Κρός για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κινηματογράφο να προσαρμοστεί στην ψηφιακή εποχή χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τρίτον να εξασφαλίσουμε ε, την ε, οικονομική αηφορία της Ευρωπαϊκής. Για το στόχο αυτό η Αντιπρόεδρος Κρός και εγώ έχουμε από κοινού καταρτήσει μια ομάδα τριών σοφών για να μας ε, συμβουλεύσουν επί του θέματος αυτού. Πέραν αυτού προσβλέπω στο να συνεργαστούμε σχετικά με την με το θέμα της ευρωπαϊκής κληρονομίας το οποίο ήδη επεξεργάζεστε και στρέφουμε τέλος εις ε, τον αθλητισμό που είναι μια ιστορική στιγμή. Με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας η Ένωση για πρώτη φορά έχει αρμοδιότητα για να βοηθήσει τη δραστηριότητα των κρατών μελών στον τομέα αυτών. Την περασμένη εβδομάδα συμμετείχα στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αθλητισμού και την άτυπη συνάντηση υπουργών και πρέπει να σας πω ότι οι προσμονές της ε, αθλητικής κίνησης είναι πάρα πολύ ψηλές η εφαρμογή των νέων διατάξεων της συνθήκης σχετικά με τον αθλητισμό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα της νέας εντολής μου και πρέπει να σας πω ότι ε, η ε, προκαταρτική δράση την οποία ψηφίσατε ήταν μεγάλη επιτυχία και θα την αναπτύξουμε περαιτέρω στο μέλλον και ελπίζω ότι θα περιληφθούν και πόροι στον προϋπολογισμό 2011. Δεύτερον, το φθινόπωρο θα σας παρουσιάσω μία ανακοίνωση για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις νέες δυνάμεις κατόπιν διαβουλεύσεως με τους ε, εμπλεκομένους και με το κοινό. Ε, το τελευταίο θέμα είναι η πολυγλωσία που ε, αναφέρεται εις την ψυχή των ευρωπαϊκών αξιών και οι γενικές διευθύνσεις μεταφράσεως και διερμηνίες αποτελούν διεθνές πρότυπο όσον αφορά την ποιότητά τους, όσον αφορά τις γλωσσικές μας πολιτικές προς τους πολίτες, πρέπει να τους βοηθήσουν να συνεννοηθούν πέραν των γλωσσικών φραγμών και να διατηρήσουν την ε, γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης. Έχουμε και ναι, άλλες γλωσσικές πολιτικές για την αφομοίωση των ε, κοινοτήτων μεταναστών και ε, την απασχόληση. Ένας άλλος τομέας είναι το θέμα των φιλολογικών μεταφράσεων ε, μέσω ε, χορηγήσεων για κινητικότητα και του χρόνου θα έχουμε τα αποτελέσματα μιας μελέτης για να ε, προχωρήσουμε στα επόμενα διαβήματα. Τέλος, δεν θέλω να σας πω πολλά περισσότερα. Αυτές είναι εν ολίγης οι προτάσεις μου για το άμεσο μέλλον και προσβλέπω στα σχόλιά σας και στην πρόθεση του διαλόγου μας. Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Είναι μεγάλο το έργο που προβλέπετε και συχνά έχω την αίσθηση ότι όλο τίτλους βλέπουμε, αλλά χανόμαστε τελικά. Ίσως ε, θα είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα εάν συνοψίζαμε κάποια πράγματα. Θα παρακαλούσα σε εσά που στέκεστε εκεί πίσω, ελάτε να καθίσετε πίσω από τις κράσινες καρτέλες. Στην ε, πέμπτη σειρά, εάν έρθουν κάποιοι συνάδελφοί μου, μπορείτε να, να παραχωρήσετε τη θέση. Δεν είναι πολύ δίκαιο αν ε, έχει έρθει κόσμος να ακούσει, να ε, στέκεται όρθιος. Εάν υπάρξει ανάγκη να παραχωρήσετε τη θέση σας, ε, φαντάζομαι θα έχετε την ευγένεια να το κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την ε, παρουσίασή σας. Προτού να δώσω το λόγο στους συναδέρφους, θα ήθελα να εκφράσω ένα πρόβλημά μου. Όλοι μας έχουμε μπροστά μας ένα έγγραφο όπου γράφει, για παράδειγμα, ε, ανακοίνωση για την απασχόληση της νεολαίας, ε, ανακοίνωση για την ε, κινητικότητα της νεολαίας, μη νομοθετικές προτάσεις. Εάν προχωρήσετε όμως στην επόμενη σελίδα, βλέπετε το, ότι το πρόγραμμα της Κομισιόν είναι το ίδιο, απλά είναι νομοθετικό. Αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό ένα εξάμεινο εργαζόμαστε σαν τρελοί πάνω σε μια ανακοίνωση και κατόπιν λαμβάνουμε νομοθετική πρόταση. Δεν είμαι βέβαια αν αυτό είναι καλό τρόπο. Ίσως θα έπρεπε από την αρχή να εργαστούμε με βάση ένα νομοθετικό πρόγραμμα για να αποφύγουμε την επικάλυψη εργασιών. Αυτή βέβαια είναι η ταπεινή μου γνώμη. Δεύτερον, ο καθένα στο μεταξύ έχει καταλάβει ότι εμένα με ενοχλεί η έκφραση youth on the move. Ε, όχι επειδή δεν είμαι υπέρ της πρωτοβουλίας αυτής, αλλά επειδή πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να καλύπτει τα πάντα. Το Youth on the Move δεν μπορεί να καλύπτει την διαβίου εκμάθηση, για παράδειγμα. Τη δεκαετία του 90 είδαμε έναν επίτροπο που ήθελε να καλύψει όλα τα προγράμματα, Εράσμους, κομμένιους κτλ. Ε, ήθελε να ε, καταργήσει όλα τα ονόματα, τα οποία όμως ε, φέρουν πολύ σημαντικό συμβολισμό και τότε το εμποδίσαμε. Τότε δεν είχαμε Youth on the Move, αλλά η διαβίω εκμάθηση μόνο εν μέρη μπορεί να ε, καλυφθεί από το Youth on the Move. Δεν μπορούμε όλα να τα καλύψουμε το πρόγραμμα αυτό, διότι η διαβίω εκμάθηση είναι ένα πρόγραμμα για ε, ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε να μην έχουμε έναν τίτλο που ακούγεται πολύ ωραίο, στον οποίο βρήκανε οι επίτροποι, ο Επίτροπος πάντων ή ε, οι άνθρωποι των δημοσίων σχέσεων πέρσι, που ουσιαστικά να καλύπτει και τη διαβίω εκμάθηση, που δεν ανήκει εκεί όμως. Ε, θα ήθελα να προ... Ε, συμβουλεύσω την Κόμισιον κατά την εκπόνηση της ε, ε ανακοίνωσης να φροντίσει το Youth on the Move να αντικαταστήσει το πρόβλημα νεολαία και να φροντίσει το πρόγραμμα νεολαία να έχει ε, καλές ε, ε, συνδέσεις με την διαβίω εκμάθηση. Αλλά όχι να, έχουμε, να τα καλύπτουμε όλα με μία μπλε σημαία με χρυσά αστέρια. Όσον αφορά την διαβίωση εκμάθηση, τα πράγματα έχουν προχωρήσει πιο γρήγορα από ό,τι πίστευα. Δεν πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να γράψουμε το Youth on the Move στην ασπίδα μας και να τα καλύπτουμε όλα. Τουλάχιστον το 60% των ανθρώπων ε, στις ε, οικονομίες μας δεν εμπίπτει εκεί. Θα παρακαλούσα λοιπόν να μην τα συγχαίουμε όλα μεταξύ τους. Ε, άλλο σημαντικό θέμα για μένα είναι ο αθλητισμός. Έχω ε, την εντύπωση, κυρία Επίτροπε, ότι πριν το 2012 δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα για τον αθλητισμό και πιστεύω ότι και η Κομισιόν φοβάται το Συμβούλιο και δεν το κάνει αυτό, διότι δεν ξέρει τι θα ε, επιτρέψει το Συμβούλιο να γίνει, διότι έχετε εδώ πέρα το πρόγραμμα για τον αθλητισμό, αλλά η Κομισιόν φοβάται μην πατήσει το πόδι κανενός άλλου και ο φόβος αυτός είναι μεγαλύτερος από την βούληση ε, να ε, εκπονήσει κάποια δράση ε, για τον αθλητισμό μέσα στα πλαίσια του προγράμματος της Λισαβόνας. περιμένετε να δείτε τι θα γίνει του χρόνου και πάλι τίποτα δεν θα γίνει. Μιλάτε για ε, παράταση του πιλωτικού προγράμματο, αλλά δεν ήταν αυτό ο στόχο. Η Κομισιόν πιστεύω έχει χρόνο και πιστεύω ότι το έχει ήδη κάνει, έχει σκεφτεί πώ μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμα αυτό. Θα ήθελα να σα παρακαλέσω να είσαστε πιο θαραλέοι, να είσαστε δραστήριοι ώστε και στον χώρο του αθλητισμού να μην έχουμε πολλά λόγια χωρίς έργα. Και ο φόβος, ξανατολμώ να το πω, είναι ο φόβος του Συμβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να είσαστε πιο θαραλέοι στην Κομισιόν. Αυτή ήταν η δική μου παρατήρηση. Δίνω τώρα το λόγο στην ε, συνάδελφο Μπατίν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ την κυρία Βασιλείου για την πληρέστατη ενημέρωσή της σχετικά με το πρόγραμμα της Κομισιόν σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που άπτονται των δικών μας αρμοδιοτήτων. Θα ήθελα να πω ότι μου δίνεται η εντύπωση πως η Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή ε, έχει συχνά ελάχιστες αρμοδιότητες. Συζητάμε για πολλά ζητήματα, αλλά οι αρμοδιότητε μας ε, είναι περιορισμένες. Θεωρώ λοιπόν πως ε, τα θέματα για τα οποία δεν έχουμε αρμοδιότητες είναι ζητήματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της ε, ατζέντα που αφορούν στους Ευρωπαίους πολίτες. Εντάξει, μπορούμε να λέμε περισσότερα ή λιγότερα πράγματα, αλλά μιλάμε πάντα για ζητήματα τα οποία αφορούν και επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Γι' αυτό θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε μια τεράστια ευθύνη και χρειάζεται να τα εμβαθύνουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Ε, μεταξύ των όσων αναφέρατε υπάρχουν δύο ζητήματα που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Το ένα αφορά το ζήτημα των πανεπιστημίων. Το η αριστεία στην ανώτατη εκπαίδευση, η κινητικότητα, η προσαρμογή των πανεπιστημιακών προγραμμάτων ε, με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουμε τους αποφύτους ε, σε, για έβρεση ναι, εργασίας κλπ. Αλλά σε πολλές χώρες όπως και στη δική μου, στην Ισπανία, ε, υπήρξαν και συνεχίζει να υπάρχει αντίδραση ενάντια στην διαδικασία της Μπολόνια και υπάρχει μια πρόταση την οποία ακούμε συχνά πυκνά ότι δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας μάλλον εμπορικεύσεις ε, του Πανεπιστημίου δηλαδή ε, θα πρέπει να προετοιμάσουμε τους νέους ε, κατά κάποιο τρόπο για να μπορέσουν να αξιάβουν εργασία. Οι νέοι αυτό το οποίο επιθυμούν είναι ναι, όντως μετά από το πέρας των πανεπιστημιακών σπουδών τους να μπορούν να βρουν μια εργασία. Αλλά τι δράσεις λοιπόν μπορούμε να αναλάβουμε προκειμένου να τους ικανοποιήσουμε τώρα. Και κάτι ακόμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι έχει ιδιαίτερη σχέση με την κρίση, ε, αφορά το ζήτημα των ε, καλλιτεχνών και όλων των, ε, των εργαζομένων στον τομέα της, του πνεύματος της διανόησης. Άκουσα ότι προτίθεστε να παρουσιάσετε μια ανακοίνωση αναφορικά με την απελευθέρωση αυτών των δικασιών και θα ήθελα εάν ε, θα μπορούσατε να μου δώσετε παραπάνω εξηγήσει αναφορικά με το πώ θα ενισχύσουμε, θα βοηθήσουμε αυτόν τον τομέα του πολιτισμού και τη βιομηχανία του πολιτισμού προκειμένου να διατηρήσουμε τις ιδιαιτερότητες μας ε, και επιπλέον να ε, τύχουν υποστήριξη για να μπορέσουν να εξέλθουν από την κρίση την οποία βιώνουμε. Ευχαριστώ. Μάκεν. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Μπορώ να είμαι σχετικά σύντομο. Ε, σίγουρα εκτιμήσαμε την παρουσίασή σα. Μα παρουσιάσατε μια ευρία γκάμα πιθανών δραστηριοτήτων. Αλλά έχω δύο ερωτήσει ε, μόνο. Ε, στον τομέα του πολιτισμού, έχετε επιλέξει τις πραγματικές σας προτεραιότητες, τα θέματα που σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και που θα υποστηρίξετε. Υπάρχει μια παροιμία, κάντε ένα πράγμα και κάντε το σωστά. Κύριε Επίτροπε, ποιο θα είναι αυτό το ένα πράγμα και η ερώτηση αυτή ισχύει και για τον αθλητισμό. Εγώ βλέπω εκεί να υπάρχει μια ευκαιρία όχι μόνο για μας ως Κοινοβούλιο ε, να δώσουμε κάποιον προσανατολισμό, αλλά και για σας βλέπουμε να υπάρχει ε, αυτή η δυνατότητα ε, ποια θα είναι η δραστηριότητα Champions League, να την πούμε έτσι, στον τομέα του αθλητισμού. Και δεν ε, αναφέρομαι σε προγράμματα του αθλητισμού που έχουν μαζική υποστήριξη ε, από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές. Ε, χρησιμοποιώ αυτή την φράση, το Champions League, για να μου πείτε, μιλάτε για τον τομέα των νέων, έχετε επιλέξει κάποια συγκεκριμένη προτεραιότητα και με την ερώτηση αυτή συνδέεται και η εξή. Πού θα χρειαστεί αυτή η μεγαλύτερη χρηματοδότηση και για τι ποσά μιλάμε. Προσωπικός μου στόχος, ε, θα ήθελα να μου πείτε ότι προσωπικός μου στόχος είναι να βρω περισσότερους πόρους για ε, ένα, δύο, τρία συγκεκριμένα προγράμματα. Μπορείτε να είσαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Θα ακούσουμε δύο ερωτήσεις ακόμα και μετά θα ακούσουμε απαντήσεις. Pani komisárka, Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σα επενέσω για τη προσπάθεια που έχετε καταβάλει και χαίρομαι που θέλετε να υποστηρίξετε του νέου. Ωστόσο, θα ήθελα να ξέρω πώ σκοπεύετε να λύσετε το θέμα τη ε, ανεργία των νέων ε, αναφέρεστε στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, ή θέλετε να ε, ε, συνεργαστείτε και με τον κοινωνικό τομέα. Όσον αφορά την ε, επαγγελματική κατάρτιση, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι νέοι δεν έχουν την αίσθηση ότι είναι καλά τα προγράμματα κατάρτισης. Από μικροί είχαν την αίσθηση ότι είναι καλύτερο να είναι κανείς δικηγόρος παρακτήστης. Η πολυγλωσσία σημαίνει πολλές γλώσσες. Αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν θα προσπαθήσει να ε, αναπτύξει την εκπάθηση γλωσσών ε, στο εγγύς μέλλον. Και επίσης πριν λίγο καιρό βρέθηκα στη Βαρκελόνη σε μία διάσκεψη και ακούσαμε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σχετικά με το γιατί απέτυχε η στρατηγική της Λισαβόνας. Μιλήσαμε για ε, την υποστήριξη της εκπαίδευσης, σε ένα πλαίσιο για την εκπαίδευση και ο καθένας που έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό γνωρίζει ότι δεν μπορούμε να πούμε στην αρχή μιας δεκαετίας ότι θέλουμε σε δέκα χρόνια να πετύχουμε τον εξή στόχο. Θα πρέπει να σκεφτούμε την όλη διαδικασία που θα μας οδηγήσει σε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε το πόσα χρόνια απαιτούνται για να αλλάξουν αυτά που συμβαίνουν. Μπορεί λοιπόν το, 2020, ε, το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 να μην είναι τόσο επιτυχές όσο αναμένουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το υποστηρίζω. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την την παρουσίασή σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τα όσα δήλωσε η κυρία Πακ, με τα σχόλια που έκανε αναφορικά με το Youth on the Move Νομίζω ότι εδώ δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ε, πτυχές ε, το διαβίου, διαβίου μάθηση παραδείγματο χάρη, διαφορά άτομα μεγαλύτερης ηλικία. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι αυτός ο τίτλος του Lifelong Learning θα έπρεπε να διαδικηθεί με τον ΑΒ τρόπο η διαβίου μάθηση. Επίσης αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι ο αθλητισμός. μου άρεσαν τα σχόλιά σας, εξάλλου παρέστην την πρώτη μέρα στην διάσκεψη της Μαδρίτης, αυτό το φόρουμ που οργανώθηκε, δεν μπόρεσα να παραμείνω για το υπόλοιπο διάστημα. Γνωρίζουμε πως οι αρμοδιότητες σε θέματα αθλητισμού ε, είναι αρμοδιότητες των κρατών μελών και σε κάποιες περιπτώσεις ε, Ισπανίας, Γερμανίας κλπ. Οι αρμοδιότητες εμπίπτουν στις ε, περιφέρειες. Θα ήταν λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό από την Κομισιό να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σε ζήτηματα αθλητισμού και να κάνει μια κίνηση συγκεκριμένη προκειμένου να δει ο κόσμος ότι έχει υπάρξει κάποια αλλαγή διότι είναι ένα ζήτημα που έχει τεράστιο αντίκτυπο στην όλη την Ευρώπη και αντίκτυπο όχι μόνο στους νέους, ιδιαίτερα στους νέους μεν διότι πιστεύουμε ότι οι νέοι που ασχολούνται με τον αθλητισμό δεν πέθουν στα ναρκωτικά ούτε στο αλκοόλ το διευκολύνει την ένταξη των μεταναστών μέσω του αθλητισμού ε, και μην μιλήσουμε τώρα για το ζήτημα υγείας, ε, του καταπολέμηση του ντόπινγκ κλπ. Εδώ με κάποια έκπληξη λέω πως αυτές οι προτάσεις που μας κάνατε και όπου αναφέρεται ο αθλητισμός δεν αποτελεί μια νομοθετική πρόταση από πλευρά σας, αλλά απλά μια ανακοίνωση ε, μια νομοθετικού περιεχομένου. Επαναλαμβάνω πως ε, θα πρέπει να κάνετε κάποια κίνηση πιο σημαντική και σας ζητώ λοιπόν κύριε Επίτροπε αυτό να αλλάξουν και να υπάρξει μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου για τον αθλητισμό για να καταδείξουμε την σημασία που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει στην, ε, στον αθλητισμό μετά από τη θέση ισχύ της συνδίκης Ευχαριστώ κύριε Επίτροπο. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με το πρόγραμμα Youth on the Move. Νεολαία και κινητικότητα. Πρέπει να ομολογήσω ότι όταν μου ζήτησε ο πρόεδρος Παρόσο να αναλάβω αυτό το ε, χαρτοφύλακα, άκουσα για το πρόγραμμα αυτό και όπως και εσείς περίμενα να δω ένα πρόγραμμα που να αφορά τους νέους και σιγά σιγά κατάλαβα ότι δεν επρόκειτο απλά για ένα πρόγραμμα, επρόκειτο για μια συνολική πολιτική και ένα πρόγραμμα ομπρέλα το οποίο θα κάλυπτε όχι μόνο προβλήματα ε, προγράμματα που αφορούν την νεολαία αλλά και την διαβίω εκμάθηση. Τι τελευταίε εβδομάδε ήμουνα και εγώ πολύ κινητική όπως ε, είπα στην πρόεδρο πριν τη συνεδρία. τι τελευταίε 16 μέρε ταξιδεύω και συνεχίζω. Αλλά ε, εκτιμώ τις ανησυχίες σας και μπορώ να πω ότι θα ήθελα καταρχήν να σα διαβεβαιώσω ότι δεν θα καταργήσουμε επιτυχή προγράμματα όπως είναι το Εράσμου, το Comenius ή το Γκρούντβι. Διότι αυτές είναι ιστορίες επιτυχίας και δεν θέλουμε να τις καταργήσουμε. Αυτό που θέλαμε όμως, αυτό που είχαμε κατά νου, ήταν να έχουμε ένα σημείο εισόδου για ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα προγράμματα αυτά, ένα σημείο που να μπορούν να λάβουν όλες τις σχετικές πληροφορίες. Θέλαμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να ε, μειώσουμε το διοικητικό άχθος. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα, αλλά σίγουρα θα εξετάσω μαζί με τις υπηρεσίες της Επιτροπής και με τον ε, Πρόεδρο ε, της Επιτροπής το θέμα αυτό, τον Πρόεδρο Μπαρόσο, ε, το θέμα αυτό και θα μεταφέρω τις ανησυχίες σας. Αυτό είχαμε εμείς κατά νου. Συγκεκριμένα δηλαδή τον Ιούνιο να έχουμε την πρώτη μας ανακοίνωση και αργότερα του χρόνου να διαμορφώσουμε το σχετικό πρόγραμμα. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά τον αθλητισμό. Θα υιοθετήσουμε ανακοίνωση για τον αθλητισμό τον Νοέμβριο. Θα υιοθετήσουμε μια προκαταρκτική δράση για τον αθλητισμό για το 2011 που είναι η τελευταία χρονιά των ε, προπαρασκευαστικών δράσεων και με βάση τις εμπειρίες που θα αποκομίσουμε από τις ε, προκατακτικές δράσεις θα υιοθετήσουμε πρόγραμμα για το 2012 και 2013. Αλλά φυσικά πρέπει να ομολογήσω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, διότι ε, στα πλαίσια των παρουσών δημοσιονομικών προοπτικών δεν έχουμε πολλά χρήματα στη διάθεσή μας για τα προγράμματα αυτά. Σίγουρα όμως θα υπάρξει πρόγραμμα για το 2012 και 2013 και κατόπιν θα οριστικοποιήσουμε το όραμά μας για το μόνιμο πρόγραμμα που θα αφορά στα χρόνια 2014 με 2020. συνάδελφος με ρώτησε σχετικά με το, το όραμά μου για τον αθλητισμό. Σίγουρα αν θέλουμε να ε, προσθέσουμε αξία σε αυτά που κάνουν τα κράτη-μέλη ή οι περιφέρειες για τον αθλητισμό θα πρέπει να τονίσουμε τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού. Οι προσωπικές μου προτεραιότητες, όπως λέτε, είναι η κοινωνική ένταξη, να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να εντάξουμε όλους τους νέους και τους μετανάστες στα πλαίσια του αθλητισμού. Ε, επίσης, ο αθλητισμός, η ε, σωματική άσκηση και η υγεία. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια του άτυπου φόρουμ όλοι ε, συμφώνησαν ότι η σωματική άσκηση και η υγεία πρέπει να είναι προτεραιότητα και επίσης ε, δίνω πολύ σημασία στην καταπολέμηση του ντόπινγκ και στην προστασία των ανηλίκων στον αθλητισμό. Αυτέ είναι οι προτεραιότητε μου. Αλλά και αθλητισμό και φύλλο είναι σημαντικό θέμα. Ε, έχουμε πολλά πράγματα να σκεφτούμε στα πλαίσια του αθλητισμού, αλλά γενικά θα έλεγα ότι δίνω προτεραιότητα στην κοινωνική πτυχή, στον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού. Επίση, θα ήθελα να τονίσω ότι για τη δική μα δουλειά πάνω στον αθλητισμό θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους ενδιαφερομένους, τους stakeholders και εννοώ όχι μόνο τις ε, μεγάλες διεθνείς και ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, εννοώ όλους τους ενδιαφερομένους. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, να δώσουμε τη δυνατότητα στον καθένα να έχει γνώμη και άποψη και να διατυπώσουμε μαζί, σε συνεργασία με αυτούς δηλαδή, ε, τι θα κάνουμε στον αθλητισμό. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι διατάξεις της συνθήκης τις οποίες θα πρέπει να σεβαστούμε και να ε, εργαστούμε πάνω στα θέματα αυτά, ε, την προστασία των ανηλίκων, ε, την κατάρτιση και την εκπαίδευση στα πλαίσια του αθλητισμού. Όλα τα θέματα αυτά είναι σημαντικά. Πολυγλωσία, τι είναι η πολυγλωσία για μένα. Δεν είναι να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να μάθει περισσότερες ξένες γλώσσες. Καλούμε τον κόσμο, καλούμε τα κράτη-μέλη να δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους νέους να μάθουν περισσότερες γλώσσες, επειδή έτσι αυτό είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο για τους νέους, για τους ανθρώπους γενικά, να επικοινωνήσουν ένας με τον άλλον. Είναι ένα μέσο ε, έβρεσης απασχόλησης. Για παράδειγμα, όταν λέμε ότι δεν υπάρχει ε, αρκετή κινητικότητα ε, στα πλαίσια της επαγγελματικής κατάρτισης, γιατί το λέμε αυτό, διότι οι άνθρωποι δεν έχουν ε, τις δεξιότητες, τα προσόντα για να είναι κινητικοί. Και ένα από αυτά τα προσόντα είναι η γνώση ξένων γλωσσών και θέλουμε να συμπεριλάβουμε τις γλώσσες, να δώσουμε τη δυνατότητα δηλαδή σε όλους τους νέους να μάθουν ξένες γλώσσες, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Ε, η ε, γλωσσομάθεια δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μια ελίτ. Βρέθηκα στη Βουδαπέστη και στη Βιέννη όταν ξανασυζητήθηκε η διαδικασία της Μπολόνια. Αναγνωρίσαμε Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμα κάποια προβλήματα με τη διαδικασία τη Μπολόνια, αλλά όλοι συμφωνήσαμε ότι είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να συνεχιστεί. Θα πρέπει να συνεχιστεί ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους φοιτητές, στους καθηγητές των πανεπιστημίων να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή. Θα πρέπει όμω επίση να συνεχίσουμε τον εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων Θα πρέπει να του δώσουμε περισσότερες δυνατότητες να είναι αυτόνομα όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, σχετικά με το διορισμό καθηγητών, σχετικά με τις προϋποθέσεις ε, για τις ε, εισαγωγικές εξετάσεις ε, των νέων, αλλά και επίσης όσον αφορά τη χρηματοδότηση, όχι μόνο από το κράτος, αλλά και από άλλες πηγές είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική η οικονομική ανεξαρτησία των πανεπιστημίων, διότι θα τα βοηθήσει να γίνουν κέντρα αριστείας, όπως θέλουμε να είναι. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι το benchmark που ξέρουμε τελικά ότι θα υιοθετηθεί από το Συμβούλιο μιλάει για τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκρίσιμη εκπαίδευση και ξέρω ότι εννοούμε εδώ και την επαγγελματική κατάρτιση. Κάποιος ανέφερε ότι μέχρι τώρα οι νέοι ε, η κυρία Ναβανταλόβα μίλησε για το θέμα αυτό. Γνωρίζουμε ότι σε πολλές χώρες, συμφωνώ μαζί σας, η ιδέα τη επαγγελματική κατάρτιση ε, δεν ε, αρέσει στου νέου, επειδή θεωρούν ότι είναι κάτι κατώτερο. Ούτε στους γονεί αρέσει και ε, περισσότερο οι γονείς επηρεάζουν τη σταδιοδρομία των νέων. Ξέρουμε όμω ότι η επαγγελματική κατάρτιση είναι πολύ σημαντική για το μέλλον μα. και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσουμε την επαγγελματική κατάρτιση, θα πρέπει να την εξυγχρονίσουμε και θα πρέπει να την κάνουμε πιο ορατή. Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια χώρα το άκουσα αυτό, ε, αλλά ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό της εικόνας της επαγγελματικής κατάρτισης είναι να την ενσωματώσουμε σε, στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, με το να μοιράζονται οι εγκαταστάσεις των πανεπιστημίων ε, θα βελτιωθεί η εικόνα της επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτή είναι μια ιδέα. Υπάρχουν πολλές ιδέες τις οποίες θα πρέπει να συζητήσουμε θα πρέπει να γίνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Η ουσία όμως παραμένει ότι στο μέλλον θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά ώστε να κάνουμε πιο ορατή ε, την επαγγελματική κατάρτιση και να την εξυγχρονίσουμε. Νομίζω ότι κάλυψα τις ερωτήσεις. Η κυρία Τρίπελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο κυρία Βασιλείου για την παρουσίασή της. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τις ιστορίες επιτυχίας, την διαβιοεκμάθηση, το Εράσμους και άλλες. Ε, δεν θα πρέπει να τα διακυβεύσουμε τα προγράμματα αυτά, ούτε να τα συμπεριλάβουμε όλα στο πρόγραμμα Youth on the Move. Είναι ε, ε, σημαντικό να υπάρχει σωστή διάκριση, διότι πολλοί πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζουν το πρόγραμμα Erasmus και ε, το πρόγραμμα για τη διαβίω και σημαντικό είναι να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό. Όταν λέτε ότι θέλετε να διευκολύνετε και να βελτιώσετε την ορατότητα, την προσβασιμότητα, σημαντικό είναι να αλλάξουμε το δημοσιονομικό κανονισμό. Όταν μιλάτε με πολίτες ή ενδιαφερομένους, ακούμε παράπονα σχετικά με το πόσο ε, δύσκολη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Υπάρχει πολλή δυσαρέσκεια ε, μεταξύ των πολιτών για τα προγράμματα αυτά και πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχοληθείτε με αυτό, διότι αλλιώς ε, θα προκαλείτε μεγάλη δυσαρέσκεια. Και φτάνω τώρα σε αυτό που είπατε για την πράσινη βίβλο. Ε, αυτά που θα συζητηθούν αύριο σχετικά με τις ε, δημιουργικές επιχειρήσεις. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ το πνεύμα της ε, σύμβασης ε, της UNESCO για την πολιτισμική ποικιλότητα. τον τομέα του πολιτισμού, πώς προβλέπετε το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι είναι σημαντικές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και με ενδιαφέρει επίσης να μάθω τι γνώμη έχετε σχετικά με μια πιθανή εναρμόνιση του copyright εντός των δικαιωμάτων ε, του δημιουργού, δηλαδή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είσαστε υπέρ, είσαστε κατά ή ε, μπορείτε να δεχτείτε κάτι τέτοιο ε, υπό ορισμένε προϋποθέσεις. Υπάρχει ήδη κάποια οριστική θέση ή εργάζεστε πάνω στη θέση σας αυτή τη στιγμή και αν ακόμα ε, το δουλεύετε το θέμα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγγνώμη κύριε Επίτροπε αν επανέρχομαι στο ζήτημα του Youth on the Move. Έλεγα λοιπόν πως επανέρχομαι στο ζήτημα του Youth on the Move διότι για να είμαι ειλικρινής δεν κατάλαβα ακόμα πως θα δομηθεί αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή τι εννοώ. Εάν θα πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά στους νέους και θα αποτελεί μια προστέμενη αξία σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα, εντάξει, το χαιρετίζουμε, με το καλό να έρθει και θεωρούμε ότι θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα για την νεολαία. Αλλά εάν αυτό πρέπει να είναι μόνο ένα δοχείο, στο οποίο όμως μπαίνουν και άλλα προγράμματα, κινδυνεύοντα παράλληλα να δημιουργήσουμε σύγχυση ή κινδυνεύοντα να περιορίσουμε οι προγράμματα τα οποία ήδη υπάρχουν, αναφέρθηκε το lifelong learning για να αναφέρω ένα, την διαβίου μάθηση, το Erasmus κλπ. Για ποιο λόγο να το κάνουμε, ποια η χρήση του, να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα δοχείο που στο τέλος ε, δεν θα έχει κανένα άλλο αποτέλεσμα από το να προκαλέσει σύγχυση με τα εφιστάμενα προγράμματα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να εμβαθύνουμε περαιτέρω αυτό το ζήτημα με τον πρόεδρο Μπαρόζο, με την Κομισιόν και εμείς ως ε, Κοινοβούλιο, αλλά κατά την άποψή μου αυτή η πτυχή που ήταν ε, εξάλλου και μία από τις πτυχές που παρουσιάστηκαν ως ιδιαίτερα καινοτόμες από τον πρόεδρο Μπαρόζο, χρειάζεται να προβληματιστούμε περαιτέρω. Και να σας ζητήσω επίσης ε, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ευρωπαϊκής πολιτικής Χρονομιάς, Αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε εμείς ε, ως Επιτροπή. Ορίστηκε ένας εισηγητής ε, και παράλληλα ισχυώδης εισηγητές, αλλά πέραν των όσων εσείς αναγγείλατε, ίσως θα μπορούσαμε να καταλάβουμε καλύτερα και αυτό θα μας βοηθούσε στις εργασίες μας σχετικά με το πώς αυτό το σήμα μπορεί να προωθηθεί, να από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των εθνικών κυβερνήσεων, δηλαδή ποια θα είναι η προσπάθεια που θα καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ευρωπή για να προωθηθούν τα διάφορες περιοχές και εγκαταστάσεις ενδιαφέροντος. Ευχαριστώ κύριε Μπόρι. Ευχαριστώ Πρόεδρε για... και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ε, ωραιότατη παρουσίαση που μας κάνατε. Ε, έτσι συμβαίνει κάθε φορά όταν ε, χτυπάει η κρίση, αυτήν ε, την ακολουθούν σε βάθος προβληματισμοί και σκέψεις και στην περίπτωση αυτή Μιλάμε για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για το 2020. Έχουμε λοιπόν φιλόδοξους στόχους, αλλά είμαστε ρεαλιστικοί. Θέλουμε να αυξήσουμε το ποσοστό των ανθρώπων με ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση στο 40%. Θέλουμε να αυξήσουμε το, τους αριθμούς, το, να μειώσουμε μάλλον τους αριθμούς των παιδιών που καταλήγουν τα σχολεία όλα αυτά είναι πολύ καλά. Αλλά τα εκπαιδευτικά μας συστήματα δεν είναι ιδιαίτερα ευέλικτα και δεν αλλάζουν από μία μέρα στην άλλη. Ε, και εξάλλου η αρμοδιότητα εμπίπτει στις ε, αρμοδιότητες των εθνικών κυβερνήσεων. Και θα πρέπει λοιπόν ε, η Κομισιόν να βρει δράσεις τις οποίες θα συντονίσει με το πλαίσιο μιας στρατηγικής. Λοιπόν, αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι φορά την βάθημα εκπαίδευση. Ακούσαμε ήδη το ζήτημα της βελτίωσης της ποιότητας αυτής της εκπαίδευσης και να την προσανατολίσουμε περισσότερο προς την αγορά εργασίας. Πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπαθειές μας στην έρευνα έτσι ώστε ο ακαδημαϊκός κόσμος να συνεργαστεί στενά με τον επιχειρηματικό. Αυτό είναι μια δυναμία του συστημάτων μας. Αυτό θα το πετύχουμε μόνο εάν εφαρμόσουμε μια μεταρρύθμιση σε βάθος, ξεκινώντας από το, ε, από το ενδιάμεσο στάδιο και καταλήγοντας ε, στον τριτογενή εκπαίδευση. Εάν ε, σκεφτούμε το πώς ο Ευρωπαίος θα ζει σε 20-30 χρόνια από σήμερα, χρειάζομαστε να προωθήσουμε τη δημιουργικότητα, την πολυγνωσία, τον αθλητισμό, τι ε, ψηφιακές δεξιότητες, ε, δεξιότητες ε, στον τομέα των επικοινωνιών και της πληροφορίας. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν και χρειάζεται τόσο εμείς ως Κοινοβούλιο αλλά και εσείς ως Κομισιόν να συντονιστούμε. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να εστιάσουμε ιδιαίτερα σε αρμοδιότητες κλειδιά και να υπάρξει μια συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις. Τώρα, σε ό,τι φορά τον αθλητισμό, πιστεύω πως θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες κλειδιά. Ήδη μας έχει απασχολήσει το παρελθόν αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να διοργανώσουμε κάποια πιλωτικά προγράμματα με την ισχύουσα ατζέντα περί αθλητισμού. Έχουμε λοιπόν κάποια περιθώρια λιγμών και αυτά θα πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Και τέλος κυρία Επίτροπε, 16 εκατομμύρια Ευρωπαίων ε, δεν έχουν τις απαραίτητες, ε, την απαραίτητη ε, κατάρτιση. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να το δούμε και αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο του Youth on the Move. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο λόγο έχει ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν ε, να επενέσω την Επίτροπο. Ε, ρώτησα κάποια πράγματα κατά την ακρόασή της ε, και μίλησε για τον αθλητισμό και χαίρομαι για αυτά που άκουσα. Δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, πανεπιστήμια τρίτου επίπεδου. Αναφερθήκατε στην στρατηγική 2020 και στην προσέγγιση των πανεπιστήμιων στην, στην επιχειρηματική κοινότητα χωρίς όμως να επηρεαστεί η αυτονομία τους. Ένα από τα προβλήματα δεν θα ήταν ότι η αυτονομία αυτή έχει οδηγήσει σε ε, σύγκριση εις βάρος των ε, ε, ευρωπαϊκών πανεπιστημίων με τα πανεπιστήμια του υπόλοιπου κόσμου. τι θα κάνετε λοιπόν για να διασφαλίσετε την αυτονομία. Και δεύτερον, ε, χάρηκα με τις ερωτήσεις ε, των συναδέλφων για τον αθλητισμό. Ε, δέχομαι και τις απαντήσεις σας. Ήδη έχετε ξεκινήσει διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Το Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα έδειξε ότι ένας από τους στόχους της στρατηγικής του 2020 που έχει να κάνει με ε, το να μένει ε, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ο κόσμος στα σχολεία, ε, ωφελεί τον αθλητισμό από το 36% των ανθρώπων που εγκαταλείπουν το σχολείο ε, στα 15 τους ε, αθλούνται, ενώ όσοι παραμένουν μέχρι τα 18 τους, ε, από αυτούς το 76% δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντική στατιστική. Και θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπε η Πρόεδρος, η Ντόρις Πακ, είπε ότι ο κόσμος περιμένει εντυπωσιακά αποτελέσματα στον αθλητισμό. Ο κόσμος περιμένει μια σαφή χειρονομία και όπως είπε ο κύριος Μάρτιν χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα τύπου Champions League. Αυτό είναι σημαντικό. Να μην καταλήξουμε να ασχολούμαστε με τι αρνητικέ πτυχές ε, του αθλητισμού όπως είναι τα προβλήματα ντόπινγκ διότι αυτό είναι περισσότερο αρμοδιότητα των κρατών μελών παρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα ήθελα, όπως είπε ο κύριος Μάρτιν, να παρουσιάσετε ένα πρόγραμμα τύπου Champions League, ώστε σε τρία-τέσσερα χρόνια ο κόσμος να πει «Α, να, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει κάτι πολύ θετικό στον τομέα του αθλητισμού». Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Well, um, I do, uh, Uh, uh, Συμφωνώ με την κυρία Τρίπελ και άλλους βουλευτές που τόνισαν τη σημασία διατήρησης προγραμμάτων όπως είναι το Εράσμους, το Κομένιους και άλλα τα οποία όλος ο κόσμος γνωρίζει. Είμαι υπέρ αυτού και ε, σίγουρα θέλω να ενθαρρύνω τη διατήρηση των προγραμμάτων αυτών. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, ε, θα πρέπει να απλοποιήσουμε τον τρόπο υποβολής ε, αιτήσεων, θα πρέπει να απλοποιήσουμε την διαχείριση των προγραμμάτων αυτών, διότι το τελευταίο τρίμηνο έχω ακούσει από τόσους ανθρώπους να μου λένε ότι εγκαταλείπουν τις προσπάθειες επειδή οι διαδικασίες είναι τόσο πολύπλοκες, που τελικά δεν κάναμε αίτηση θα πρέπει να διευκολύνουμε τον κόσμο και γι' αυτό, εάν θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι όσον αφορά την κινητικότητα, θα πρέπει να διευκολύνουμε την υποβολή αιτήσεων ε, στα προγράμματα κινητικότητας. Ε, και θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα για κινητικότητα όχι μόνο στους φοιτητές των πανεπιστημίων και στα παιδιά των λυκείων ή στους ε, δασκάλους, στους καθηγητές, αλλά και στους πιο νέους. Συγγνώμη, στους νέους εργαζομένους, θα πρέπει, σε αυτούς που λαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση, θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα αυτή της εμπειρία στους ανθρώπους αυτούς, να εργαστούν δηλαδή ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είχα τη δυνατότητα στην Ισπανία να συναντηθώ με κάποιες ομάδες νέων που συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα ανταλλαγών και βλέπει κανείς τα ωφέλη. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα αυτή σε όλους τους νέους. Να σας πω λίγα λόγια για τον πολιτισμό και τις ε, δημιουργικές επιχειρήσεις. Στις μελέτες μας βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές πολιτισμού και δημιουργικότητας αποτελούν πηγή διατήρησης ε, του πολιτισμικού πλούτου της ε, κοινωνίας της Ευρώπης. Ταυτόχρονα συμβάλλουν σημαντικά στις οικονομίες μας. Εντυπωσιάστηκα όταν είδα τα νούμερα. Κάποιες πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης είχαν τεράστιο εισόδημα από την απόκτηση του τίτλου, διότι κατάφεραν να μετατρέψουν τις, κοινωνίες, τις κοινότητες τους από βιομηχανικές σε πολιτισμικές, μάλλον να δώσουν αυτή την πολιτιστική εικόνα στις κοινωνίες του Η Γλασκόβη, το Λίτζ, η Λίλ, το Έσεν ίσως ε, να έχει τα, ε, το ίδιο αποτέλεσμα. Σημαντικό είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις αυτές, τις ε, πολιτιστικές ε, και ε, δημιουργικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Όπως σας είπα, πρόκειται για διπλή επιτυχία, διότι αφενός έχουμε αυτή την πολιτιστική έκφραση και όταν μιλάμε για, για δημιουργικές επιχειρήσεις, μιλάμε για τα βιβλία που διαβάζουμε, τη μουσική που ακούμε, τι ταινίε που βλέπουμε. Μιλάμε για πολλούς διαφορετικούς τομείς, τους οποίους θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Και όπως σας είπα, αύριο θα υιοθετήσουμε πράσινη βίβλο για τις ε, επιχειρήσεις στον τομέα του πολιτισμού, για να ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να τις υποστηρίξουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η ευρωπαϊκή πολιτιστική ετικέτα. Βλέπουμε, πιστεύουμε ότι θα έχει ωφέλη και Είχαμε αίτημα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο η διακυβερνητική πρωτοβουλία αυτή να γίνει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Νομίζω ότι το όφελος της πρωτοβουλίας αυτής θα είναι ότι θα δώσουμε μια ε, αίσθηση ιδιοκτησία στον Ευρωπαϊκό Πολιτή, μια ε, αίσθηση πατρίδας ε, πολιτισμού, διότι τα διότι τα μνημεία που θα συμπεριληφθούν δεν είναι τα παραδοσιακά μνημεία κλασικής ομορφιάς. Έχουμε τα μνημεία ε, του ε, ε, πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλάμε για διαφορετική πρωτοβουλία. Και τέλος, Θα συνενώσουμε τα μνημεία που θα λάβουν αυτή την ετικέτα και θα δούμε πώς μπορούμε να τα κάνουμε πιο ορατά στους πολίτες. Και δεν μιλάμε μόνο για αυτά μνημεία, αλλά και για άλλα. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία έχουμε το διάταγμα του 1867 για την κατάργηση της θενατικής ποινής. Ε, αυτό θα έχει την ετικέτα αυτή, διότι αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ε, έτσι θέλουμε να προσθέσουμε αξία με την ετικέτα αυτή στην ουσία. Όσον αφορά τα πανεπιστήμια, θέλουμε να προωθήσουμε την αριστεία. εκπονούμε μελέτη σχετικά με την ιεράρχηση των πανεπιστημίων, διότι πιστεύουμε, την αξιολόγηση των πανεπιστημίων, διότι πιστεύουμε ότι οι φοιτητέ δεν λαμβάνουν εμπεριστατωμένε αποφάσει ε, όσον αφορά την ιεραρχία των πανεπιστημίων, την αξιολόγηση των πανεπιστημίων. Ε, ελπίζουμε η μελέτη αυτή να είναι έτοιμη του χρόνου για να δούμε Πώ μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να έχουμε μια σφαιρική αξιολόγηση των πανεπιστημίων, η οποία να διαφέρει από την παραδοσιακή ιεράρχηση της ε, Σανγκάη, ανάλογα με την κατεύθυνση και το όραμα του κάθε πανεπιστημίου, διότι ε, αυτή τη στιγμή συγκρίνουμε άνισα πράγματα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα τεχνικό πανεπιστήμιο ένα πολυτεχνείο δηλαδή, με ένα ε, πανεπιστήμιο ανθρωπιστικών σπουδών. Θα πρέπει να έχουμε διαφορετικές κατηγορίες για τα πανεπιστήμια, ώστε ο φοιτητή ή ο νέος να μπορεί να κάνει εμπεριστατωμένη επιλογή του εκπαιδευτικού προγράμματος που θέλει να παρακολουθήσει. Και μια συμπληρωματική παρατήρηση για τον αθλητισμό. Ήμουνα πριν επίτροπος για την υγεία και με βάση τις εμπειρίες μου από εκεί θέλω να δώσω δυναμική στον αθλητισμό για όλες τις ηλικίες. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να ασκούνται, να αθλούνται. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους αλλά και των σπουδών τους και μετά το πτυχίο να συνεχίσουν να αθλούνται. Και στην τρίτη ηλικία, ακόμα και οι, οι ηλικιωμένοι πρέπει να συνεχίσουν να αθλούνται, διότι έτσι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την υγεία ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες αυτές είναι οι φιλοδοξίες μου, να προωθήσουμε δηλαδή τον αθλητισμό από πολύ μικρή σε μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία. Όσον αφορά την ιδέα του να έχουμε ένα πρόγραμμα τύπου Champions League, θα έχουμε τη δυνατότητα να το εξετάσουμε αυτό. Όλες οι ιδέες σχετικά με την κοινωνική πτυχή, τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού, Και όταν μιλάμε για το πρόγραμμα 2012-2013 και για το μέλλον γενικά, ακούμε τις, ε, ε, τις θέσεις σας και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε ένα πρόγραμμα ναυαρχίδα, να το πούμε έτσι, το οποίο θα προσθέσει ευρωπαϊκή αξία στις δράσεις των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Έχω ακόμα πέντε συναδέλφους. Ε, μας μένουν μόνο 15 λεπτά. Σας παρακαλώ λοιπόν, φροντίστε όλοι να μην θέσετε τις ίδιες ερωτήσεις που ήδη ακούσαμε. Ένα μισή λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Κύρια Βασιλείου, καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα σχετικά με τον αθλητισμό και τις ε, πολιτιστικές επιχειρήσεις. Θα επικεντρωθώ όμως περισσότερο σε αυτό που δεν συζητήθηκε πολύ, την πολυγλωσία. Έχει πολλές πτυχές το θέμα αυτό που συζητώνται εντός των κρατών μελών. Μιλάμε για τους νέους που μαθαίνουν γλώσσες άλλες από τη μητρική τους. Ε, εσείς αναφερθήκατε στις κοινότητες των μεταναστών, οι οποίες όμως ε, αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για πολλά κράτη-μέλη. Ε, μιλάμε για άτομα όχι απαραίτητα από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από χώρες Εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλούν τη δική του γλώσσα. Πώ θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Εισέρχεται κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μιλάει άλλε γλώσσε και γι' αυτό δεν έχει ίσες ευκαιρίες, δεν μπορούν να προχωρήσουν στη ζωή του με τον τρόπο που μπορούν άνθρωποι που δεν προέρχεται από μεταναστευτικέ κοινότητε. Υπάρχει λοιπόν εδώ σημαντικό θέμα κοινωνική συνοχή και κινητικότητα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε, τι προτείνετε να γίνει. Ευχαριστώ κύριε Καμαϊβέτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ε, διατυπώσατε ε, φιλόδοξες, φιλόδοξους στόχους, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης. Αναφερθήκατε στα πανεπιστήμια, στην επαγγελματική κατάρτιση, ε, στην προβληματική των ανθρώπων, στο πρόβλημα των ανθρώπων που εγκαταλείπουν το σχολείο στην εκπαιδευτική πολιτική έχουμε το ιδιαίτερο πρόβλημα που δεν έχουμε σε άλλους τομείς, ότι όλοι εδώ πέρα πρέπει να ακολουθήσουμε την επικουρικότητα. Και οι δηλώσει του κυρίου Μπαρόσο οδήγησαν στα γερμανικά κρατήδια σε σημαντικέ ε, αντιδράσει, διότι στον τομέα τη ευρωπαϊκή πολιτική ακούστηκε δεν έχει η Ευρώπη λόγο. Οι στόχοι μας μπορούν να επιτευχθούν ε, όχι μόνο με πολλά ωραία προγράμματα, τα οποία είναι σίγουρα είναι καλά και θα πρέπει να εφαρμοστούν. Ε, αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς, θα πρέπει να ε, έχουμε πιο στενή συνεργασία και διατύπωση κοινών στόχων που να τηρήσουν όλα τα κράτη-μέλη, να δεσμευτούν όλα τα κράτη-μέλη ε, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να πετύχουν όλου του στόχου αυτού. Εσεί ω Επίτροπο, ε, ενδεχομένω σε συνεργασία μαζί με εμά ε, στο Κοινοβούλιο, ε, τι δυνατότητε ε, βλέπετε να υπάρχουν για συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για κοινού στόχου. Ε, ώστε πέρα από τα προγράμματα στον τομέα του πολιτισμού να μπορέσουμε στην Ευρώπη να προοδεύσουμε. Rova ε, Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την προσέγγιση της. Ο ενθουσιασμός με τον οποίο αδράξατε θα το ζήτημα είναι κάτι το ιδιαίτερα θετικό και ελπίζω να μπορέσετε για να μπορέσουμε από κοινού να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τώρα σχετικά με το πρόγραμμα του 2020 ελπίζω να μπορέσει να προχωρήσει και να υλοποιηθεί. Βεστος, εμείς δεν ε, είχαμε αναμεχθεί σε αυτό το ζήτημα ιδιαίτερα αυτή εξ αρχή. Ε, τώρα το θέμα είναι πώς ε, θα μπορέσει να υπάρξει κατάλληλο συντονισμό ε, με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να έχουμε μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Και κάτι ακόμα το οποίο εθίγει αφορά στα πανεπιστήμια. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια όπως η Oxford και το Cambridge, ε, είναι ανάμεσα στα 20 καλύτερα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους ε, για να αναβαθμίσουμε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και να τα καταστήσουμε πιο ελκυστικά έτσι ώστε οι νέοι μας ε, να μην αναχωρούν και να μεταβαίνουν στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε το επίπεδο της ποιότητας των πανεπιστήμιων μας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπεναράμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, κυρία Βασιλείου, για την παρουσίασή σας, την οποία βρήκα ιδιαίτερα φιλόδοξη. Αναβαρθήκατε στην πολυγλωσία και να σας πω και εγώ την απόψή μου. Κάτε με, η γλώσσα δεν είναι μόνο ένα μέσο επικοινωνίας, κάθε γλώσσα φέρει έναν κόσμο μαζί της και έναν πολιτισμό. Αυτό σημαίνει ότι το να ευνοήσουμε τις γλώσσες θα μας δοθεί μια δυνατότητα να έχουμε μια ευρύτερη πρόσβαση στον ε, κόσμο. Αυτό είναι απαραίτητο στον τόσο περίπλοκο κόσμο στον οποίο ζούμε. Επανέρχομαι τώρα στο ζήτημα των φοιτητών. Είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο να επιθυμούμε το 40% των νέων να μπορούν ε, να ε, περνάνε στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Το ζήτημα είναι αφορά τους ε, φοιτητές ε, από τα χαμηλότερα κοινωνικά επίπεδα. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουν αυτοί οι φοιτητές να έχουν δυνατότητα να, ε, να φοιτήσουν. Προτίθεται λοιπόν να προτείνεται ένα καθεστώς, ένα καταστατικό των φοιτητών ανάλογα με το οικονομικό τους επίπεδο. Σε ό,τι φορά τώρα το θέμα της απασχόλησης, το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, εντάξει καλές είναι σπουδές, αλλά και μετά θα πρέπει να είναι σε θέση να εξέχουν εργασία οι απόφοιτοι τώρα. Ειδικά με την έκθεση ΒΕΡ, να σας πω κατά πόσον εξετάσατε την δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα και στον τομέα της εκπαίδευσης. Πόσες ε, θέσεις απασχόλησης θα μπορούσαν να, δημιουργηθούν με τη στρατηγική προτείνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα ό,τι είπατε για την, για την πράσινη βίβλο. Καταρχήν θα έπρεπε πρώτα να το διαβάσει κανείς, αλλά έχω μία παράπλευρη ερώτηση, ερώτηση. Διότι πρέπει να βρούμε ταλέντα και να τα εκπαιδεύσουμε και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε θαυμάσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά ελάχιστους εξαίρετους καλλιτέχνες, διότι διάφορα πράγματα έχουν αλλάξει τα τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό σας κάνω την ερώτηση χωρίς να είμαι βέβαιος ότι μπορείτε να μου απαντήσετε διότι πάντοτε μου έλεγαν αν, αν θέλεις να γίνεις σκηνοθέτη στο Πότσνταμ ε, ε, ε, ή εκεί, για να γίνεις κάμεραμαν εδώ ή εκεί. Τώρα όμως μπορεί να πω ότι ίσως αυτά που θα σου έλεγα πολλές... αλλά ε, οπωσδήποτε στο Βερολίνο, διότι εκεί υπάρχουν ναι μεν ε, ε, ασταθείς συνθήκες εργασίας, αλλά εξαιρετική και ειδική με κομπιούτερ. Υπάρχει ένα πολιτιστικό περιβάλλον το οποίο έχει μεγάλη σημασία για να αναπτυχθούν τα ταλέντα και έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ότι έχει καλύτερη εκπαίδευση για τους καλλιτέχνες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα τελευταία απάντηση της κυρίας Βασιλείου. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με τον κύριο Μπίσκι δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημά σας. Μπορώ όμως να εκφράσω την ε, ε, θεωρία μου και το όραμά μου, διότι όταν μιλάμε ε, για ταλέντα, θέλουμε να δώσουμε εις τους νέους τη δυνατότητα και την ευκαιρία να με τον τρόπο με τον οποίο αυτοί φαντάζονται, δηλαδή εκεί που έχουν κάποια κλίση, διότι προς το παρόν περιορίζουμε πάρα πολύ τους φοιτητές μας. Από πολλοί νέους τους δίνουμε μία πολύ περιοριστική κατεύθυνση ενώ θα έπρεπε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να διερευνήσουν και άλλα θέματα. Τον πολιτισμό, τον αθλητισμό ή άλλες κλήσεις τις οποίες μπορεί να έχουν, άλλα ταλέντα μπορεί να έχουν. Πώς λοιπόν θα δώσουμε ουσία στο όραμα αυτό. Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν μπορώ να σας απαντήσω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Σύμφωνο ότι η πολυγλωσία δεν είναι μόνο ένα εργαλείο, είναι και μία πολιτιστική έκφραση, είναι ε, μέλος του πλούτου μας ε, ο πλούτος της Ευρώπης είναι η πολυγλωσία και εκτός από τις 23 επίσημες γλώσσες έχουμε περίπου 60 άλλες γλώσσες τις οποίες στηρίζουμε διότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον πλούτο και στην πολυμορφία η οποία υπάρχει, ποικιλομορφία που υπάρχει στην Ευρώπη. Το να μάθει κανείς μία γλώσσα είναι ένα θέμα αλλά η διατήρηση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας είναι κάτι τελείως διαφορετικό και εξίσου σημαντικό. Για να έρθω στην κυρία Χάνιμπολ και να πούμε πώς μπορούμε να διατηρήσουμε αυτές τις κοινωνίες. Καταρχήν θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα ή μάλλον να τις ενθαρρύνουν να μάθουν τη γλώσσα της χώρας που τους φιλοξενεί. Μόνο έτσι θα ενταχθούν στην κοινωνία και συγχρόνως πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα και την ενθάρρυνση να διατηρήσουν την μητρική τους γλώσσα. Δεν το πίστευα, αλλά στο Φιγκαρό διάβασα ότι υπάρχουν 600 γλώσσες οι οποίες μιλούνται στην Ευρώπη. Τόσο πολύμορφη, πολυμορφική είναι η κοινωνία στην Ευρώπη. Λοιπόν, ε, ε, μέσω των διαρθρωτικών ταμείων μέσω ίσως ε, του κοινωνικού προγράμματος θα μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε την περιφέρεια, την τοπική αυτοδιοίκηση να διοργανώσει μαθήματα για αυτούς τους λαούς για να διατηρήσουν την γλωσσική τους πολυμορφία. Όσον αφορά την ε, ε, εξοικείωση με τη γλώσσα της χώρας που τους φιλοξενεί πρέπει να είναι προτεραιότητα για να μπορέσουμε ε, να επιτύχουμε φέτος που είναι η χρονιά της καταπολέμησης της, ε, του κοινωνικού αποκλεισμού. Τώρα, πώς θα προωθήσουμε την στρατηγική της Λισαβόνας και τη στρατηγική της Ευρώπης του 2020. Στη στρατηγική της Λισαβόνας είχαμε θέσει πάρα πολλούς στόχους. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε αναφέρει περίπου 20 διαφορετικούς στόχους. Και δεν ακολουθήσαμε ακριβώς τι γινόταν κάθε χρόνο. Οπότε στο τέλος διαπιστώσαμε ότι δεν επιτύχαμε τους στόχους αυτούς. Συμφωνώ λοιπόν με αυτούς οι οποίοι λένε ότι πρέπει να περιορίσουμε τώρα τους στόχους τους οποίους θα καταρτήσουμε και να καταρτήσουμε μόνο 20 ε, και μόνο πέντε με συγχωρείτε και ε, να ε, προσπαθήσουμε όχι να ξεμπροστιάσουμε αυτούς που δεν πάνε καλά αλλά να εντοπίσουμε τις δυσκολίες ε, που, αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη και πώς θα επιτύχουν τους στόχους αυτούς, πώς δηλαδή θα αντεπεξέλθουν των δυσκολιών. Όταν λοιπόν μιλάμε για στόχους, η, αυτή είναι η ε, ευρωπαϊκή μέση όρη όταν μιλάμε για την εγκατάλειψη του σχολείου. Το ποσοστό δεν είναι το ίδιο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει λοιπόν να δούμε πού πάει καλά κάποιο κράτος, πού έχει δυσκολίες, πού έχει αδυναμίες και με ποια προγράμματα μπορούμε να τους βοηθήσουμε να επιλύσουν τις δυσκολίες τους. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της στρατηγικής Λισαβόνας και της στρατηγικής του 2020. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι πιο αισιόδοξη. Δηλαδή πιστεύω ότι συνεργαζόμενοι και είπα ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να ε, μπορέσουμε ε, να καταρτήσουμε σωστούς εθνικούς στόχους. Πρέπει πέραν των εθνικών στόχων να συνεργαστούμε, να δούμε πώς θα συνεργαστούμε και πώς θα τους βοηθήσουμε να επιτύχουν στους στόχους που, τους οποίους μόνοι τους έχουν θέσει. Αυτά είχα να σας πω κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Βασιλείου. Ήθελα να θυμηθούμε όλοι ότι πολλά ελέγχθησαν. Δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά όπως αντιλαμβάνεστε. Ακόμη και αν τα συζητάμε, ακόμη και αν τα επεξεργαζόμαστε πολλά πράγματα θα γίνουν στις χώρες μας και αν δείτε πόσο καταρτίστηκε η ε, στρατηγική της Μπολόνια ε, τότε λυπάμαι διότι δεν είμαι τόσο αισιόδοξη για το μέλλον ε, θα πρέπει όχι να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, αλλά να κάνουμε κάτι νέο και επικοδομητικό. Έχω να σας πω όμως κάτι για το Youth on the Move, για την ε, νεολαία εγκινήση. Μην το χρησιμοποιήσετε σαν λόγο για να πείτε ότι διευκολύνουμε τη διαδικασία, διότι με αυτή την κίνηση δεν θα απλοποιήσετε τίποτα. Αν ε, εμείς ζητάμε να απλοποιήσουμε το Comenius ε, τα πάντα, για χρόνια, από όταν υπάρχει ο κανονισμός. Ορισμένα κάναμε, ορισμένους μικρούς στόχους επιτύχαμε, αλλά ε, όλα βασίζονται ε, στο δημοσιονομικό κανονισμό και θα πρέπει ε, να το μειώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί διαφορετικά ο κόσμος θα βαρεθεί τα προγράμματά μας. Η νεολαία εγκινήσει δεν πρόκειται να βελτιώσει τα πράγματα ή να μειώσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Να το έχετε στο μυαλό σας. Χρειαζόμαστε τη διαβίου μάθηση ως έχει τώρα. Χρειαζόμαστε την νεολαία εγκινήση που χρησιμοποιεί ένα μέρος της διαβίου μάθησης αλλά θα πρέπει να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε το πρόγραμμά μας γιατί ε, πρέπει ε, να βοηθήσουμε και τους πολίτες οι οποίοι έχουν συνηθίσει τώρα τα προγράμματα της διαβίου μάθησης που έχουν επιτύχει. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι δύο ωραίες ημέρες στην ε, Κίνα και σας ευχαριστώ που ήρθατε να μας μιλήσετε. Υφυπουργό. Take a seat. should use your phones because I speak in German. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, Λοιπόν, τώρα θα προχωρήσουμε στο εμερίσιο, στην ημερήσια διάταξή μας. Ο Υφυπουργό Αθλητισμού της Ισπανίας μας είχε ζητήσει να μας παρουσιάσει εδώ τις δραστηριότητες στον τομέα του αθλητισμού της Ισπανικής Προεδρίας. Στο 8, στο κανάλι 8 είναι τα ισπανικά. Χαιρόμαστε λοιπόν που ο Γενικός Γραμματέας, αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, ο Χαϊμέλη Σαβέσκι που το όνομά του βέβαια είναι μάλλον πολωνέζικο και όχι ισπανικό, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι η Ευρώπη έχει αφομοιωθεί τόσο πολύ, ώστε να έχουμε έναν εκπρόσωπο της Ισπανικής Προεδρίας, Χαϊμέλη Λισαβέτσκι. Και θα μας μιλήσει για τις ισπανικές δραστηριότητες. Ξέρουμε ότι το φόρουμ αθλητισμού στη Μαδρίτη εμποδίστηκε από το νέφος της στάχτης του ηφαιστείου και εγώ είχα ε, μία συνάντηση όπου δεν μπόρεσα να μεταβώ αλλά ελπίζουμε ότι τώρα η Ισπανική Προεδρία μπόρεσε να θέσει τις βάσεις της εργασίας την οποία περιέγραψε η κυρία Βασιλείου. Έκανα προηγουμένως μία παρατήρηση ότι φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, είναι και τόσο επιμελής στην πολιτική αθλητισμού διότι φοβάται το Συμβούλιο ότι το Συμβούλιο δεν θέλει να κάνει για τον αθλητισμό αυτό που εμείς ζητούμε βάσει της επικουρικότητος. Μπορείτε ίσως να καθησυχάσετε αυτές τις ανησυχίες μας και να μας πείτε τι προβλέπετε και τι έχετε σκεφτεί στην Ισπανική Προεδρία και παρακαλώ τώρα ακόμη και ο Αντιπρόεδρος να μπορέσει να μας μιλήσει. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον αναπληρωτή Υπουργό. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για τα γενικά σας λόγια. Αποτελεί ιδιαίτερη ικανοποίηση για μένα, αλλά και τιμή συνάμα να βρίσκομαι εδώ ενώπιον της Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω προκειμένου μετά να υποβληθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός ερωτήσεων. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στο πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Θα ονόμαζα ένα πλαίσιο μεγάλων προσδοκιών, διότι οι προσδοκίε προέρχονται από την έγκριση τη Δίκη Λισαβόνα, όπου αναγνωρίζεται ο αθλητισμό ω αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για τι ιδιαιτερότητε του τομέα και αναφέρει ότι θα πρέπει να προάγουμε τον αθλητισμό Λέει επίσης ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την ισότητα και το άνοιγμα στον αθλητισμό και στους αγώνες. Ε, επίσης αναφέρει η συνθήκη ότι χρειάζεται να προάγουμε την συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με διεθνείς ε, αθλητικές οργανώσεις ε, και ομοσπονδίες και επίσης ε, αναφέρονται και, αναφέρεται και το ζήτημα των συστάσεων. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν προσπάθησε να πράξει η Ισπανία κατά τη διάρκεια αυτού του τετράμινου τη Προεδρία τη. Δεν ξεκινάμε όμω το 0, δεν ξέρω είναι το 0, διότι ήδη από το 1991 προετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ανακοίνωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αθλητισμό, μια ε, κήρυξη του Άμστερνταμ το 1997 για τις μη οικονομικές πτυχές που άπτονται με τον αθλητισμό, την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις εκθέσεις Μπελέν Μαυρομάτη και κάποιε άλλες πτυχές. Επίσης υπήρξε λευκή βίβλος για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό το 2007 με ένα πρόγραμμα δράση ε, με 23 δράσεις και επίσης υπήρξαν δράσεις που αφορούσαν την οικονομική πτυχή του αθλητισμού και απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, απόφαση Μπόσμαν 1985 95 ε, ε, ε, και ως εκ τούτου καταλαβαίνετε ότι δεν ξεκινήσαμε από το μηδέν. Έχουν γίνει διάφορες συνεδριάσεις άτυπες υπευθύνων, υπουργών, γενικών γραμματέων, αθλητισμού κλπ. με την Ευρωπαϊκή Τροπή και φυσικά υπήρξε κάποια σημαντική πρόοδος οι οποίε ε, θα συμπεριληφθούν σε αυτή τη λευκή βίβλο. Τώρα, αυτή την βασική στιγμή, θα πρέπει να καθορίσουν κάποιε προτεραιότητες και χρειάζεται να λάβουμε υπόψη αυτή η κοινωνική και όχι μόνο οικονομική πτυχή του αθλητισμού. Οι προτεραιότητες ε, που έχουμε καταδείξει μέσω του, του τρίου τη Προεδρίας και στη εργασία των κρατών μελών και της Κομισιόν είναι πέντε. Πρώτα απ' όλα κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού. Δεύτερον, η προαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων και αθλητικών δραστηριοτήτων για την βελτίωση τη υγεία των πολιτών. Τρίτον, κοινή καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό και η εκπαιδευτική και η διδακτική ε, του αθλητισμού και κάτι ακόμα ε, στενή συνεργασία με του διεθνεί αρμόδιους Οργανισμού και ομοσπονδίας ε, ε, μέσω ενός δομημένου διαλόγου, δηλαδή ενός μόνιμου διαλόγου ανάμεσα στα αθλητικά κινήματα και τις δημόσιες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη και το θέμα του κοινωνικού διαλόγου. Για να ολοκληρώσω αυτές τις σκέψεις, ε, θα θέλω να πω ότι έγινε μια συνάντηση των Γενικών Διευθυντών τον ε, Φεβρουάριο στην Ισπανία και επίσης μια πρώτη συνεδρίαση έγινε την 1η Απριλίου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τροπή και για τον ρόλο για το αθλητισμό στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε και η Πρόεδρος, το ε, ζήτημα της εφιστιογενούς ε, τέφρας δεν, μπορεί, μας, δεν μας βοήθησε στην διεξαγωγή αυτής της συνεδρίασης. Έγινε όμως η συνεδρία 20-21 Απριλίου των Υπουργών στην Μαδρίτη και κάτι ακόμα, ένα συνέδριο των Υπουργών που θα διεξαχθεί προς τα τέλη Μαΐου στις Βρυξέλλες, Υπουργών του Αθλητισμού φυσικά. Και θέλουμε να ολοκληρώσουμε την Προεδρία μας ε, με μια ενδιαφέρουσα πτυχία, ένα ευρωπαϊκό συμπόσιο για τον αθλητισμό που θα οργανωθεί τον Ιούνιο. άκουσα μπαίνοντα ότι η Κομισιόν ε, ετοιμάζει ένα σχέδιο ανακοινώσει, ε, το οποίο προτίθεται να υποβάλει στο Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί κατά τη διάρκεια της προσεχούς ε, Βελικής Προεδρίας και έτσι θα αποκρισταλώσουμε κάποιες πτυχές τις οποίες προαναφέρθηκαν. Τώρα συγκεκριμένε ισπανικές προτάσεις ήταν πρώτον δημιουργία μιας νέας ομάδας εργασίας για το θέμα των ίσων ευκαιριών και της κοινωνική ένταξης των αθλητισμού. Βρισκόμαστε στο έτος για την καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού. θα εκδώσουμε κάποιες νόμες που θα εφαρμόσουν εκ των τα κράτη-μέλη και δεύτερον να ενισχυθεί ο δομημένος διάλογος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι αυτό μπορεί να έχει, υπάρχουν κάποιες διαφορές ή κάποια σύγκρουση από ε, απόψεων. Οι στόχοι μπορεί να είναι οι ίδιοι, αλλά εμείς εδώ προθούμε να συντονίσουμε τις ε, θέσεις ε, του καθενός και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια συμβουλευτική επιτροπή μόνιμου χαρακτήρα. Στην ενδρία στον Βρυξελών θα μιλήσουμε για τη συνθήκη τη Λισαβόνα και τι απόψει όλων των κρατών αλλά και του Συμβούλου και τη Κομισιόν και θα Και τώρα από πλευρά δημοσίων αρχών θα πω ότι θα είναι παρόν τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Το Κοινοβούλιο γι' αυτό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Τώρα, ο Εμείς δεν πρέπει φυσικά να προσδιορίσουμε ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι των ε, κρατών μελών. Ε, να υπενθυμίσω, Πρόεδρε, αν μου το επιτρέπετε, στο ζήτημα της ε, από αποβίωσης ε, του κ. Σάμαρανκ. Ε, λυπούμεθα για την ε, θάνατό του. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτές τις συνεδριάσεις να συμμετέχει και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αλλά και επίσης κάποιες ομοσπονδίες. Εντάξει, θα πρέπει να βρούμε λοιπόν σύνθεση, αλλά θα πρέπει κατά βάθο ε, αθλητικοί παράγοντες να συμμετέχουν σε αυτά τις συζητήσεις. Χρειάζεται λοιπόν ε, να συμπεριληφθεί αυτή η έννοια του διαλόγου σε όλες τις δράσεις, θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδης σημασία και υπάρχει και μια άλλη συνεδρίαση αυτή του ομάδας ε, που σας προανέφερα στις 10 ε, Μαΐου μαζί με την ε, συνεδρίαση των ε, αρμοδίων υπουργών Χρειάζεται φυσικά να υπάρξουν συνεδριάσεις θεματικές βραχυπρόθεσμα, μεσοπράθεσμα για να δούμε τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε είχε υποθεί μία ιδέα, είχε, γίνει, είχε υπάρξει μάλλον μία ιδέα σχετικά με το ζήτημα αυτό, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, από ό,τι ξέρω στον ανακοίνωση υπάρχει κάποια αναφορά στον αθλητισμό για το 2012-2013 και ολοκληρώνω, επιτρέψτε μου να πω τα εξής πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη έλεγα, ε, ε, κοινοτική ηγεσία στα θέματα αθλητισμού. Τι εννοώ, εννοώ ότι θα πρέπει ομαδικά να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε και να βαδίσουμε, να μην είμαστε λοιπόν μόνο θεατές των τεχνομένων Πρέπει να είμαστε λοιπόν ε, πιο προορατικοί Το κείμενο, μάλλον η έκθεση του Κοινοβουλίου θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική ε, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την αφοσίωσή σας, η οποία φάνηκε και από την ταχύτητα με την οποία εκφωνήσατε την ομιλία σας. Έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε καλά αποτελέσματα, αλλά προέρχομαι από μια χώρα από όπου κοιτάμε με επιφύλαξη τα θέματα αυτά. Υπάρχουν θέματα που θεωρούμε ότι δεν αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να ξέρω τι αντίκτυπο βρίσκουν τα λόγια σας στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν χώρες που δεν θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα, υπάρχουν κάποιοι που είναι τελείως κατά, υπάρχουν κάποιοι που με ενθουσιασμό ε, θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτά. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Μπέλετ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ε, εκτίμηση για τις φιλοδοξίες της Προεδρίας. Ε, κυρία Πακ, ε, συμμερίζομαι τη θέση σας και την ερώτησή σας για το θέμα αυτό και έχω και μία συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Υφυπουργέ, που έχει να κάνει με την ισορροπία στον αθλητισμό, ένα ερώτημα κρίσιμο για το μέλλον του αθλητισμού στην Ευρώπη. Η αλληλεγγύη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με βάση την εξισορροπημένη ανακατανομή δικαιωμάτων τηλεόρασης που αποτελούν το βασικό εισόδημα για όλους τους τομείς του αθλητισμού και ιδιαίτερα για το ποδόσφαιρο που είναι το πιο δημοφιλέ άθλημα στην Ευρώπη. Και επαναλαμβάνω αυτά που ήδη είπατε κυρία Πρόεδρε, ε, δεν είναι στόχο τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ούτε με τη συνθήκη τη Λισαβόνα να ρυθμίσουμε τον αθλητικό τομέα. Αυτό ε, είναι. Ε, αυτό είναι θέμα των αρμοδίων αρχών, αλλά πρέπει να σπρώξουμε τη FIFA, την UEFA και τις εθνικές αρχές προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όλα τα σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλα τα μέλη της UEFA τα ε, δικαιώματα ε, ε, τηλεόρασης πολλούνται μαζικά. Εκτός από την Ισπανία και η Ιταλία του χρόνου θα ε, θα περάσει στο ε, σύστημα ε, ομαδικής πώληση. Στην Ισπανία όμως έχουμε μεμονωμένες πωλήσει των δικαιωμάτων. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η θέση σας για το θέμα αυτό και τι επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί στο θέμα αυτό, διότι η πρώτη κατηγορία μαζί με την πρώτη αγγλική κατηγορία, την πρώτη κατηγορία στην Γερμανία αποτελούν κατηγορίες με τους με τα πιο επιτυχή πρωταθλήματα στον κόσμο και μπορούν να αποτελέσουν και πρότυπο, πράγμα που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ερώτηση λοιπόν, μπορείτε να ε, επηρεάσετε την πολύ σημαντική αυτή διαδικασία και πιστεύω ότι τώρα είναι η σωστή στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο. Έχετε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως ε, και σε άλλα κράτη-μέλη, όπως και σε άλλες κατηγορίες, ε, Κάποιε ε, κορυφαίες ομάδες τη Ισπανία αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Είναι λοιπόν ώρα για δράση, είναι κατάλληλη στιγμή. Η Ισπανία είναι μια χώρα ποδοσφαιρική και την τελευταία φορά που πήγα στη Βαρκελόνη παίζαν στο πρωτάθλημα. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω μια σοβαρή ερώτηση. Είναι πολύ καλό που είσαστε ανοιχτός στη συζήτηση αλλά εγώ δεν είμαι ειδική και πρέπει να σας ρωτήσω πώς μπορείτε ε, να ε, εκπροσωπήσετε όλους το, τα σπορ διότι πλέον ε, του, ε, του ποδοσφαίρου υπάρχει το curling, υπάρχει το σκάκι ε, και θα ήθελα να ξέρω πώς εσείς επιλύετε αυτή τη δυσκολία, πώς την αντιμετωπίζετε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ε, για τον αθλητισμό και θα θέλαμε και εμείς να είχαμε θέσεις για το προοδοσφαιρικό πρωτάθλημα την του Αφρική και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο μέλλον. Η κυρία Μπαντία. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον ε, αναπληρωτή Υπουργό κύριο Λασεύσκη μολονότι μας έκανε κάποιες ε, παρατηρήσεις αλλά σε ιδιαίτερη υψηλή ταχύτητα όπως είπε και η Πρόεδρος ε, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της κοινωνικής ένταξης που και εσείς στήξατε. Νομίζω ότι τα αθλητικά, η αθλητισμό συγγνώμη, ως μπορεί να αποτέλεσε ένα στοιχείο κοινωνικού ε, κοινωνική ένταξη. ιδιαίτερα έχοντα κατά νου του μετανάστες αλλά και του νέου. Γνωρίζετε αναφίβολα καλύτερα από μένα το ζήτημα, έχετε εμπειρίε θετικέ που διεξάγονται σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία οι αρμοδιότητε που η συνθήκη τη Λισαβόνα παρέχει στον Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα αθλητισμού θα μπορούσαν να βελτιώσουν, να επηρεάσουν ε, τον συντονισμό ανάμεσα στις πρωτοβουλίες και της εμπειρίας βέλτιστων πρακτικών που ήδη φύστανται για την κοινωνική ένταξη και για την ενσωμάτωση επαναλαμβάνω των μεταναστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να χρησιμεύσουν ε, για να ε, υπάρξει κάποιο κανόνα ο οποίο θα ακολουθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν εάν εντός αυτών των προτεραιοτήτων για την κοινωνική ένταξη προβλέπονται κάποιε πρωτοβουλίε ή σκέφτεστε να προωθήσετε συγκεκριμένε πρωτοβουλίε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και στη δικιά μου χώρα δεν θα παριστάμαστε εις ε, το πρωτάθλημα αλλά θα οργανώσουμε το πρωτάθλημα του 2012. Θέλω να κάνω μία ερώτηση κύριε Υπουργέ. Παρουσιάστε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο σημειώνει ότι οι ε, διατάξεις συνθήκες της Λισαβόνας ε, θα εφαρμοστούν από το Συμβούλιο Υπουργών και από τους Υπουργούς. Μία ερώτηση. Η μόνιμη συμβουλευτική ομάδα για τον αθλητισμό την οποία εισάγατε εδώ για πρώτη φορά έχει φιλόδοξους στόχους και μάλιστα συγκεκριμένες αρμοδιότητες κλειδιά. Τώρα οι νέοι θα πρέπει να αποκτήσουν και ορισμένες ε, δεξιότητες ε, κλειδιά για τον αθλητισμό, γιατί θα τους είναι χρήσιμες στη ζωή τους περαιτέρω. Ε, έχετε χρησιμοποιήσει αυτή την πτυχή στις στρατηγικές αθλητισμού των κρατών μελών και δεν έχει κάθε κράτος μια τέτοια στρατηγική και αν δεν υπάρχει ενιαία εφαρμογή δεν θα χρειαστούν αυτές οι αρμοδιότητες. Πιστεύετε ότι θα ήταν σκόπιμο να βελτιώσουμε το σύστημα εκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως μεταξύ κρατών μελών όπου υπάρχουν διαφορετικές εμπειρίες. Θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ των υπουργών που είναι υπεύθυνοι για τον αθλητισμό για να βελτιώσουν τις δεξιότητες των ανθρώπων που ασχολούνται στο επιμορφωτικό πρόγραμμα διότι δεν ικανοποιητικό αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Κέλλη από την Ιρλανδία. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ένα προερώτημα. Αναφερθήκατε ε, στο θέμα ότι ε, ο αθλητισμός θα έχει σωστή εκπροσώπηση. Τι γίνεται ε, για τις ε, οργανώσεις που εκπροσωπούν τον αθλητισμό. Αυτές πώς θα εκπροσωπηθούν στο όργανο αυτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον αναπληρωτή Υπουργό, διότι κατέδειξε ότι γνωρίζει σε βάθος το ζήτημα και έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Θα ήθελα μεταφέρει αυτόν τον ενθουσιασμό και προς την ε, Κομισιόν και να προωθήσει αυτούς τους κανόνες του οποίους ανέφερε. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπε η κυρία Μπαδία για την σημασία του αθλητισμού ως ε, σύστημα για την ε, κοινωνική ένταξη και την άθληση των νέων μας. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις, παραδείγματος χάρη, στο θέμα του ντόπινγκ. Νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι η επικάλυψη νομοθεσίας Έχουμε την αθλητική νομοθεσία και τις κυρώσεις που βλέπει όταν ένας αθλητής ε, το πάρεται και όπως και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, υπάρχει, στο, υπάρχει το δίκαιο, το δικαίωμα μάλλον προσφυγή στα εθνικά δικαστήρια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιμηκύνει τις προθεσμίες, τις διορίες κλπ. Και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Τώρα μιλήσαμε και για το θέμα της κατανομής των πόρων για τον αθλητισμό. Θα ήθελα να κάνετε κάποιο σχόλιο αναφορικά με το σύστημα τον ε, προπό των στοιχημάτων που υπάρχουν και την ε, κατανομή αυτών των εσόδων και κατά πόσον ε, περνάνε και σε άλλα αθλήματα πέραν του ποδοσφαίρου αυτά τα κοντήλια. και κάτι ακόμα. Ε, υπάρχει δυνατότητα σε ό,τι φορά το ποδόσφαιρο να περιοριστούν αυτά τα υπέρογγα χρήματα τα οποία δίνονται στους ε, ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες υπερβολές και αυτό οδηγεί κάποια προβλήματα στις ε, αθλητικές ομοσπονδίες ε, κλπ. Και κάτι ακόμα, το ζήτημα της οργάνωσης των αθλητικών δραστηριοτήτων στα στις πόλεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πείτε στην Κομισιόν αυτή η πρόταση, η μη νομοθετική, υποβάλει, υποβάλλει, να μετατραπεί σε νομοθετική πρόταση. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, μακρηγόρησα. Και η τελευταία ερώτηση είναι από την κυρία Καμαέβατ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Η μία μου ερώτηση έχει σχέση με αυτά που είπε τώρα ο κύριος Μπέλετ το θέμα της κεντρικής εμπορίας διότι ακούω από τους γερμανικούς ομίλους ότι θα θέλαν να έχουν μια ευρωπαϊκή νομοθεσία επί του θέματος που θα διευκρινίζει ότι ε, η κεντρική αυτή ρύθμιση δεν θα συγκρούεται με το ευρωπαϊκό ε, δίκαιο ανταγωνισμού. Μπορεί να υπάρξει μια διευκρίνηση επ' αυτού του θέματος και δεύτερον παρακαλούμε να μας στηρίξετε στις επόμενες συζητήσεις προϋπολογισμού γιατί ε, πέρυσι με τα λύπης διαπιστώσαμε ότι τα μέτρα τα οποία είχε προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον προϋπολογισμό ε, είχαν περικοπεί πάρα πολύ κατά μισό εκατομμύριο ε, προσπαθήσαμε να τα αυξήσουμε αλλά δεν επιτύχαμε την αύξηση η οποία έφτανε στο επίπεδο του προηγουμένου έτους. Εάν λοιπόν θέλουμε να προχωρήσουμε πέραν των προκαταρτικών μέτρων, δηλαδή για να επανέλθω σε αυτά που είπατε στην αρχή της συζητήσεώς μας σήμερα το πρωί, θα πρέπει επί ευρωπαϊκού επίπεδου να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε όλα τα θετικά στοιχεία στον προϋπολογισμό και γι' αυτό πιστεύω ότι η Ισπανική Προεδρία θα πρέπει και στα θέματα του προϋπολογισμού και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού να αποτελέσει ένα σύμμαχό μας επί του θέματος. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο Γενικός Γραμματέας τώρα έχει συγκεντρώσει αρκετές ερωτήσεις στις οποίες μπορεί να απαντήσει και του δίνω το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Ναι, πριν ε, μιλούσα πολύ γρήγορα γιατί μου είχαν πει ότι αν ε, πάρεις πολύ χρόνο τότε θα υπάρξει χρόνο να σου θέσουν ερωτήσεις. Ζητώ συγγνώμη, το συγγνώμη από τους διερμηνείς ε, για την ταχύτητα με την οποία μίλησα. Τώρα να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις που μου θέσατε, ξεκινώντας από την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Μπελέτη, ο οποίος μίλησε για το θέμα των ε, τηλεοπτικών δικαιωμάτων αναμετάδοσης ε, εγώ ε, δεν ήθελα να μιλήσω για τη χώρα μου, αλλά θα μιλήσω. Θέλω να σας πω ποιες είναι οι προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου λοιπόν νομίζω ότι αυτό το οποίο εσείς λέτε αφορά και άλλα κράτη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίε στο ζήτημα αθλητισμού. Αν με ρωτάτε τη γνώμη, τη γνώμη μου βασίζεται στην Λευκή Βίβλο, βρίσκεται εδώ, είναι μια γνώμη υπέρ της ε, αλληλεγγύης. Είναι διαφορετικό ότι στη Λευκή Βίβλο γίνεται ένας προβληματισμός σχετικά με τα δικαιώματα αυτά, τα οποία θα πρέπει να είναι κατά πόσο ατομικά ή συλλογικά. Αυτό που έχει σημασία ε, δεν, έχει, δεν είναι το πώς θα έχουν αυτά τα δικαιώματα, είναι συλλογικά ή αν θα είναι ομαδικά ή ατομικά, αλλά θα πρέπει να βασίζονται στο κριτήριο της ελληνικής. Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα, κάτι ακόμα. Στην Ισπανία δουλεύουμε και στην Βουλή υπάρχει μια υποεπιτροπή που συγκεκριμένα αύριο θα ψηφίσει ε, κάποια ψηφίσματα και δουλεύουμε για την ε, υποβολή ενός ε, νόμου για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Σε, αυτό τον επαγγελματικό, σε αυτή την νομοθεσία θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος θα ασκεί έναν οικονομικό έλεγχο να μην υπάρχουν ε, ανισορροπίες ανάμεσα στα έσοδα και τα έξοδα. Θα Κοιτάξουμε λοιπόν να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα και φυσικά πολλές άλλες πτυχές. Πιστεύω ότι αυτή είναι καλή στιγμή για να προχωρήσουμε στην μεταρρύθμιση του, του επαγγελματικού αθλητισμού και κάτι ακόμα χαιρετίζω την πρωτοβουλία της UEFA και ο κύριος Πλατινής συγκεκριμένα που δεν αφορούν μόνο τα ζητήματα κοινωνικού διαλόγου, αλλά και το ζήτημα του οικονομικού fair play. Θέλω να πιστεύω ότι χρειάζεται, χρειάζονται αυτά τα κριτήρια και αυτές οι ομάδες που έχουν ε, κάποια οικονομικά προβλήματα να μην μπορούν να συμμετέχουν στις αθλητικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θετικό ζήτημα. Τώρα, σε σχέση με το τι θα μπορούν να κάνουν η FIFA και η UEFA αναφορικά με την πώληση των δικαιωμάτων να πω ότι συμφορώ με αυτά που δηλώσατε και να πω και κάτι. Πιστεύω, εγώ δεν είμαι νομικός, είμαι επιστήμονας, είμαι ερευνητής. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια ευρωπαϊκή εναρμόνιση σε αυτό το ζήτημα. Τα κρατημέλη πρέπει να λαμβάνουν τι αποφάσει του. Αλλά προσθέτω κάτι ακόμα. Μια που μιλήσατε για την Ισπανία, δεν υπάρχει ένα νόμο, ένα κανόνα, ένα, μια νομοθεσία που να απαγορεύει την, ε, το θέμα τη ε, και να ρυθμίζει το ζήτημα αυτών των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει, υπάρχει απόλυτη ελευθερία, υπάρχει αυτονομία, υπάρχει ελευθερία. σχετικά με το πώς θα απολυθούν αυτά τα δικαιώματα, ε, ατομικά, μεμονωμένα δηλαδή ή ομαδικά. Υπάρχει, όπως είπα, ελευθερία τώρα. Είναι υποχρέωση του, του δημοσίου να δημιουργήσει μηχανισμούς αλληλεγγύης πέρα τη νομικής πτυχής αυτής κατά αυτή. Συμφωνώ λοιπόν με τα λεγόμενά σας. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και την συνεργασία σας στο Κοινοβούλιο, διότι είχα την ευκαιρία να διαβάσω την έκθεσή σας. Και χαίρομαι που μπορώ και σας συναντώ. Και με τώρα μια άλλη ερώτηση που τέθηκε. Το θέμα της εκπροσώπησης ε, των αθλητών. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα σύστημα όπου υπάρχουν διεθνείς νομοσπονδίες ε, που είναι και όλες αυτές οι αντιπροσωπείες ε, έχουν ε, την ε, βαρύτητά τους σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο. Δεν πρόκειται να ε, βρούμε ένα νέο σύστημα και δεν ξέρω αν πόσε είναι αυτέ οι ομοσπονδίε, αν είναι 60-70 σε παγκόσμιο επίπεδο, πάντω το σύστημα όσο έχει λειτουργεί αποτελεσματικά. Φυσικά οι πιο ισχυροί έχουν δυνατότητε να κάνουν περισσότερα πράγματα από άλλου που έχουν λιγότερα, είναι λιγότερο ισχυροί και οικονομικά. Δεν νομίζω λοιπόν πως υπάρχει κάποια αντιφατικότητα από το να με το να συσταθεί μια ομάδα συντονιστική η οποία θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε διότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στην συμμεσχύουσα κατάσταση και την συνεργασία με τις υπόλοιπες ομοσπονδίες είτε αυτές είναι μικρές είτε μεγάλες. Νομίζω λοιπόν ότι οι ομοσπονδίες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και, για ρόλο και σε επίπεδο διαπαιδαγώγησης αλλά και εκγύμνασης θα λέγαμε των αθλητών. Λοιπόν αυτή η Συμβουλευτική Επιτροπή και σε συνεργασία με τις ομοσπονδίες θα δουν πώς θα μπορέσουν να συνεργαστούν. Νομίζω ότι θα υπάρξει συμμετοχή των ε, εμπλεκομένων αναφίβολα. Ε, σας ευχαριστώ κύριε μου για την παρέμβασή σας ε, διότι ό,τι αφορά τις βέλτιστες πρακτικές, την βελτίωση του συντονισμού, ανταλλαγή πληροφοριών, θα είναι ευπρόσδεκτο έτσι αναφέρεται στην ανακοίνωση, στο σχέδιο ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως εκ τούτου πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση ε, με τις ευκαιρίες για να απαντήσω σε ένα άλλο ερώτημα που έχει σχέση με τον περιορισμό των ε, αμοιβών ε, που είπες φίλε μου. Νομίζω ότι η έννοια του αθλητισμού στην Ευρώπη διαφέρει από αυτήν των Πολιτειών. Στις Πολιτείες θεωρείται ότι είναι ε, μια βιομηχανία αναψυχής ε, διασκέδασης ε, στην ε, Ευρώπη είναι τα πράγματα διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ευρώπη Είπατε ότι είσαι φιλελεύθερος, δεν μπορεί να υπάρχει δυνατότητα περιορισμού των αμοιβών, αλλά Θα ήθελα να μιλήσω τώρα για την Ισπανία και να πω ότι δαπανάται μόνο το 70% των εσόδων το πολύ σε ό,τι αφορά μισθού κλπ. Άρα μπορούμε να κάνουμε και κάποιε συμφωνίε και να μην περιορίζουμε τι αμοιβέ αλλά τις, τις, ε, τα ποσά που ε, χορηγούνται για την πληρωμή των αμοιβών. Υπάρχει λοιπόν ένα ανώτατο όριο, ένα χ% Τώρα, κύριε Μπόρις, ε, καλή τύχη σε ό,τι φορά την διοργάνωση αυτού του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι θα είναι ε, πολύ καλό πρωτάθλημα. Τώρα, για τη συμβουλευτική ομάδα, ποιες ε, θα είναι οι βασικές αρμοδιότητες. Θα πρέπει να προσδιοριστούν. Κάναμε μια αρχική πρόταση στην συνεδρίαση των Γενικών Διευθυντών και αυτό το οποίο ζητήσαμε είναι ότι σύμφωνα με αυτά που θα εγκρίνει η Βελική Προεδρία τους προσεχείς μήνες, αυτή η ομάδα η οποία θα έχει συσταθεί θα πρέπει να αναφερθεί στη σύνθεσή της, την ατζέντα της κλπ. κλπ. Εάν έχει... Θα πρέπει να έχει λοιπόν κάποια σαφή αρμοδιότητα για να μπορέσει να προωθηθεί ο διάλογος δεν θα πρέπει να υπάρξουν τώρα ε, κάποιες διαφωνίες και διαφορές που θα εκδηλωθούν μέσω του τύπου, αλλά θα πρέπει αυτές οι διαφορές ακόμα και αν υπάρχουν να λιανθούν, να περιοριστούν. Ε, Δίχως το διάλογο, αν κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί. Και εντός έξι μηνών θα πρέπει να υπάρξει μια συνεδρίαση για να ρυθμιστούν όλα τα προβλήματα. Επίσης, εάν ε, δεν υπάρχουν νομοθετικές αρμοδιότητες, ε, να πω το εξής, εάν 27 κράτη-μέλη συμφωνήσουν, τότε αυτή η συμφωνία, αυτή η άποψη θα έχει τεράστια, τεράστιες επιπτώσεις, τεράστιο αντίκτυπο. Μπορούν λοιπόν να συμφωνήσουν ε, οι ομοσπονδίες για να επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος. Ή τι άλλο όλα αυτά θα είναι ενδιαφέροντα. Τώρα, σχετικά με τη βελτίωση τώρα του συντονισμού και την ε, εκπαίδευση στα κρατη Νομίζω ότι και ο Σαντιακοφίδης έκανε την ίδια ερώτηση. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αναφέρεται στο σχέδιο ανακοίνωσης. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και συμφωνώ με την γνώμη που εκφράσατε. Κάτι ακόμα σχετικά με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, το μη επαγγελματικό και την εκπροσώπησή του σε αυτή την ομάδα. Κοιτάξτε, ε, υπάρχει ε, μια ε, αίτηση να ακουστούν ε, τα γνώμες των ομαδικών αθλημάτων. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για τον επαγγελματικό κόσμο, αλλά μιλάμε και για τους αραστέχνες, για τον αραστέχνισμό. Εγώ θέλω λοιπόν να υπάρχει εκπροσώπηση όλων των πλευρών. Στην Μαδρίτη εκπροσωπήθηκαν ε, από την ΔΟΕ, τη Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών. Εντάξει, ο κ. δεν μπόρεσε να παραστεί, αλλά ήταν ο επικεφαλής της Ισπανικής ΔΟΕ, ε, κάποιων ευρωπαϊκών κρατών ε, ΔΟΕ εκπροσωπήθηκαν, ε, ομοσπονδίας, άθλητες κλπ. Υπήρχαν ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, που δεν... Όλο αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και να προσπαθήσουμε να εκπροσωπηθούν ο μεγαλύτερο αριθμός ε, τόμων. Θα πρέπει λοιπόν η πληροφορία να ρέει. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να υπάρξει ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός εισαγωγικών με όλους τους εκπροσώπους των αθλητικών οργανώσεων, ομίλων, διών κλπ. Συλλόγων και ό,τι άλλο θέλετε. Κύριε Φίσα, το ζήτημα του ντόπινγκ, ναι, εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν ε, να πετύχουμε την εναρμόνιση σε επίπεδο νομοθεσιών σε κάποιες χώρες θεωρείται αδίκημα η διακίνηση, η κατοχή, το να επιβάλλει σε κάποιον αθλητή να χρησιμοποιήσει αυτές τις ουσίες και λοιπά και ο νέος κώδικας που έχουμε τώρα στην Ισπανία αλλά και στη Γαλλία. Δεν θέλω να επισέλθω τώρα σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, η ανταρμόνιση είναι κάτι το δύσκολο. Αλλά στην συνεδρίαση που είχαμε, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε για και να πάμε πέρα από αυτές τις ε, συμφωνίες με την Ιντερπόλ, με τα τελωνία, με τα εργαστήρια κλπ. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό ε, και έχει φυσικά και την ε, ποινική πτυχή του. Τώρα, υπάρχει όμως και η άλλη συζήτηση που αφορά τις ε, οργανώσεις και τις ομοσπονδίες κάθε χώρας. Ένας αθλητής μπορεί να προσφύγει σε ένα αθλητικό δικαστήριο. Ε, αυτό όμως δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με ε, ένα ψήφισμα το οποίο θα ζητάει να γίνονται πιο γρήγορα οι όλες οι διαδικασίες και, να μην, και οι διορίες να είναι οι αυτές. Όλα αυτά είναι προβλήματα. Τώρα για το ντόπινγκ να σας πω ότι προηγούμενα όταν αναφέρθηκα στην διάθεση όλων και τη γνώμη όλων, ότι δηλαδή πρόκειται για μια μάστιγα κλπ. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον, έχουμε τον ε, οργανισμό, διεθνή οργανισμό κατά του ντόπινγκ, εγώ συμμετέχω σε αυτόν, ε, επιστήμονας και θεωρώ ότι αυτός ε, ο οργανισμός είναι θεμελιώδης, ουσιώδης, διότι εξετάζονται όλες οι πτυχές. Επίσης το θέμα της προστασίας δεδομένων είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Στην... Ε, πρόσφατα λύσαμε ένα πρόβλημα, αλλά ξέρουμε ότι το ζήτημα είναι περίπλοκο. Αναφερθήκατε στο ζήτημα των ε, αμοιβών, εντάξει απάντησα, τώρα ε, ο μειογένεια των ε, τίτλων. Ε, συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Εγώ δεν είμαι μόνο απλά αναπληρωτής ε, μιας χώρας, υπουργός που, μιας χώρας που έχει την ε, Προεδρία, αλλά θεωρώ ότι η Κομισιόν έκανε με εξαιρετική εργασία. Πρόκειται για μια πολύ καλή ανακοίνωση τώρα, αλλά δυστυχώς έχουμε την οικονομική κρίση και αν φυσικά μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε, τότε θα έχουμε έναν ε, προϋπολογισμό ικανό για αυτό το θέμα που μας απασχολεί. Έχουμε αρμοδιότητες, θα έχουμε και ένα πρόγραμμα για δραστηριότητες. Τώρα, πόσα θα μπορέσουμε να ε, βάλουμε σε αυτό το κονδύλι για τη βελτίωση της υγείας, την καταπολέμηση του ντόπινγκ κλπ. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις ε, εγώ το, αυτό, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα το προσπαθήσω. Και τελευταία παρέμβαση. Στο πρώτο τμήμα της. Δεν την κατάλαβα απόλυτα. Αν μπορείτε να το διευκρινίσετε περαιτέρω το πρώτο τμήμα της ερώτησής σας. Τώρα για την ε, πολιτική του προϋπολογισμού, κοιτάξτε, οποιοδήποτε αρμόδιος ε, για κάποιο ζήτημα, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ζητάει όλο και περισσότερα χρήματα. Εγώ το λέω στον ε, Πρωθυπουργό Θαπατέρο, αλλά τι να κάνουμε υπάρχουν περιορισμοί, αλλά φυσικά έχουμε τώρα περισσότερες αρμοδιότητες και έτσι μπορούμε να αγωνιστούμε προκειμένου να αποκτήσουμε και περισσότερα κονδύλια. Ευχαριστώ. Gracias. Ευχαριστώ πολύ. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι κάποιος μπορεί να μιλήσει πιο γρήγορα και από μένα αλλά βλέπετε πάντοτε διαψεύδομαι. Ήταν πολύ, πολύ χρήσιμο με πολλές πληροφορίες και ελπίζω ότι και στο μέλλον με την ε, βοήθειά σας ε, ε, στην Βελγική Προεδρία ο Ιβο Μπέλετ θα πιέσει να υπάρχει ένας σοβαρός υπουργό στο θέμα αυτό ε, και εφόσον θέλει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το, η τωρινή Προεδρία του Συμβουλίου θέλει, το Κοινοβούλιο επίσης επιθυμεί, άρα τι άλλο χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτά που μας επιτρέπει τώρα η συνθήκη. Σας ευχαριστώ και πάλι και καλή σας τύχη.